E Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, καθίστε. Λέει η Πρόεδρος. Και να αρχίσουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Καλωσορίσατε όλοι και ιδίω να καλωσορίσουμε τους προσκεκλημένους μας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και να καλοδεχτούμε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Αντιπρόεδρο, την κυρία Ρέντινγκ. Η κυρία Ρέντινγκ ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη σημερινή συνάντηση. Ε, είναι συνδιοργάνωση επομένως ε, Κομισιόν και Κοινοβουλίου Θα τις δώσω ευθύς αμέσως το λόγο της κυρίας Αντιπροέδρου, ούτω ώστε να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Σα Σας ευχαριστώ κυρία Ματσόνη, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω σε αυτό το σεμινάριο το οποίο πιστεύω θα σταθεί πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες όπως γνωρίζετε η νέα συνθήκη της Λισαβόνας έχει αποτελέσει μια πραγματική επανάσταση γιατί στο επίκεντρο των πάντων όλων των πολιτικών μας έχει βάλει τον πολίτη. Και αυτός ο χάρτης των δικαιωμάτων έχει αποκτήσει πλέον δεσμευτική σημασία. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο χάρτης θα πρέπει να αποτελεί τον μπούσουλα, μια επεξίδα τον μπούσουλα για πάσα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τα κρατημέλη, ούτως ώστε ε, θα πρέπει τα κρατημέλη έτσι να επαγρυπνούν για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Αποτελεί την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτός ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τις βασικές μας ελευθερίες και δικαιώματα. Αυτό το έχουμε συλλάβει ως ένα μέσο ε, ούτως ώστε όλοι να απολαύουν αυτόν τον θεμελιών δικαιωμάτων υπό πάσα περίσταση ε, από ό,τι ρυθμίζεται από το κοινωτικό δίκαιο, πρόκειται για ένα ζωντανό νομοθέτημα που κάθε μέρα ωφελεί. Κάθε μέρα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και από τα δικαστήρια που έρχεται η ώρα να εφαρμόσει το κοινωτικό δίκαιο. Και το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επομένω ενέκρινε τη στρατηγική που θα αφορά την ε, υιοθέτηση αυτού του χάρτη και ο στόχος είναι ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτό αφορά όχι μόνο όσους ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη των κρατών μελών και επίσης να υπάρχει ε, και εμπιστοσύνη πλευρά του κόσμου, του κοινού για τις πολιτικές μας, ε, για τον τρόπο υλοποίησης και εφαρμογής αυτών. Οι προτεραιότητές μας είναι το να γίνεται σεβαστός αυτός ο χάρτης, παντού από κάθε νομοθέτη. Και Εμεί με τη σειρά μα, όταν προετοιμάζουμε κάποιε προτάσει, να λαμβάνει την υπόψη κάποιε τροπολογίε Συμβουλίου και ε, Κοινοβουλίου και αυτό να φτάνει μέχρι την ημέρα κατά την οποία οι προτάσει αυτέ γίνονται δίκαιο. Δίκαιο το οποίο καλούνται να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη και βεβαίω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεμπνεί και ελέγχει τα κράτη-μέλη. Επομένω, θα πρέπει να ισχύει αυτό, να ισχύει αυτό ο χάρτη να γίνεται σεβαστό. Οπότε ε, ο κόσμο έχει συγκεκριμένε προσδοκίε όσον αφορά τη θέση εφαρμογή αυτού του χάρτη. Και έχουμε πει στην ετήσια έκθεση του Μαρτίου για φέτο, όσον αφορά τον χάρτη. Με αυτή την έκθεση θέλουμε να παρακολουθήσουμε την πρόοδο της εφαρμογής του χάρτη και επίσης έτσι να παρασχεθούν πληροφορίες σε σχέση με το τι γίνεται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεσμικών οργάνων, κρατών μελών, ούτως ώστε να εφαρμοστεί ο χάρτης. Αυτό τώρα το οποίο σας ενδιαφέρον είναι να μπορούμε να δούμε το πόσες επιστολές έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ζωντανό ενδιαφέρον από πλευρά του κόσμου. Όμω, υπάρχει και ένα πρόβλημα, διότι τα τρία τέταρτα αυτών των επιστολών αφορούν ζητήματα και περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το κοινωτικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει επομένω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση για τον σκοπό του χάρτη αλλά και της αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όντως, ξέρετε κι εσείς ότι δεν ισχύει για τα πάντα αυτός ο χάρτης και αφορά μόνο την περίπτωση κατά την οποία κάποιο κράτος μέλος καλείται να εφαρμόσει το κοινωτικό δίκαιο διότι ο χάρτης δεν δίνει μια γενική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο ώστε να παρέμβει σε περίπτωση παραβίασης θεμελιωτών δικαιωμάτων. Ακριβώς αυτό είναι το σημείο στο οποίο και για το οποίο υπάρχει η παρεξήγηση. Αυτή η παρεξήγηση επομένως ε, είναι αντικείμενο μελέτης από πλευρά του Ευρωπαίου μεσολαβητή, διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τον οποίο 72% των Ευρωπαίων δεν θεωρούν ότι έχουν πλήρως και δεόντως ενημερωθεί για τον χάρτη. Κυρίε και κύριοι, αυτό είναι ένα από του λόγου για του οποίου σήμερα μαζευτήκαμε εδώ. Διότι Συμφωνούμε όλοι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Και θα πρέπει να αποφύγουμε την ε, απογοήτευση από πλευράς όλων. Θα πρέπει επομένω όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια και όλα τα θεσμικά όργανα τόσο να ενημερώσουμε του πολίτε για το πότε ισχύει και πότε δεν ισχύει ε, αυτό ο χάρτη. Πρόκειται για μια κοινή μα ευθύνη. Ε, και όταν λέω ε, κοινή ευθύνη εννοώ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και υπηρεσίες και επίσης την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, αλλά, αλλά ενώ εδώ ότι είναι ευθύνη και των κρατών μελών. Η δέτηση έκθεση του 2010 για την εφαρμογή του χάρτη είναι το πρώτο βήμα. Αυτό το βήμα το έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να ενημερώσει τους πολίτες επ' αυτού και αυτό τονίζει τα συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία έχουν ε, να αντιμετωπίζουν τα φυσικά πρόσωπα και κατά αυτόν τον τρόπο εξηγείται γιατί μερικές φορές δεν μπορεί να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λόγω αυτών των ε, ορίων που έχει τάξει συνθήκη στις αρμοδιότητές της. Είναι όμως κατά τη γνώμη πάρα πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι ακόμα και αν αυτός ο χάρτης δεν ισχύει ε, σε σχέση με αυτά τα οποία κάνουν Ευρωπαϊκέ υπηρεσίε και όργανα σε μερικέ περιπτώσει. Τα δικαιώματα συνεχίζουν και αποτελούν αντικείμενο εγγύηση σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό δυνάμει των εθνικών συνταγμάτων. Άρα δεν υπάρχει εδώ κάποιο κενό. Απλώ, αντί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σκητάλη την παίρνει κάποιο άλλο. Οπότε πρέπει όμως να είναι ενημερωμένοι και οι συμπολίτε μας το ότι τη σκητάλη την παίρνει κάποιος άλλος από τα ευρωπαϊκά όργανα. Και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ περίπλοκο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να, να υπάρχει επικοινωνία σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί ακριβώς αυτά τα θέματα είναι περίπλοκα και είμαι βεβαία ότι ακριβώς τα ίδια ισχύουν και σε εθνικό επίπεδο. Επομένως, είναι σημαντικό και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο να μπορέσουμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Να δούμε τι θα κάνουμε αυτά τα προβλήματα. Να δούμε με ποιο μέσο, με ποιο εργαλείο θα ενεργούμε σε κάθε περίπτωση μια που οι πολίτες τυψούν να λάβουν μια απάντηση. Επόμενος, τι να κάνουμε, τι να βελτιώσουμε. Οι πολίτες και οι συμπολίτες προσδοκούν κάποιους μηχανισμούς επανόρθωσης οι οποίοι να είναι επαρκείς, να είναι προσβάσιμο τόσο ώστε να λυθούν τα προβλήματα αυτά και δεν τους καίγεται δεν, δεν, δεν δίνουν δεκάρα για αυτά τα οποία ε, ονομάζουν οι νομικοί πηγή δικαίου διότι αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος είναι να υπάρχει κάποιο είδους αποτελεσματική στήριξη ε, αρρωγή όσον αφορά τα δικαιώματά τους και χρειάζεται επομένως ενημέρωση ενημέρωση και να υπάρχουν επίση και κάποια μέσα, 11 εξώδικα, Επανόρθωση και αυτό το οποίο χρειάζεται και θα πρέπει επομένω να γίνουν τα κατάλληλα διαβήματα τόσο ώστε η κατάσταση αυτή να αποκατασταθεί και επίση να υπάρχει ενημέρωση σε σχέση με το πού θα παραπονεθεί, πού θα καταγγείλει κανεί την παραβίαση των θεμελιώδων δικαιωμάτων. Α, έχουμε και αυτό το, το, το, την διαδικτυακή πύλη, πόρταλ, ε, παύλα, justice, τη δικαιοσύνη. Να λοιπόν, σήμερα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Θα πρέπει να κάτσουμε εδώ και θα πρέπει να τεθεί στο τραπέζι το πώ μπορούμε να συνεργαστούμε, πώ θα διερευνήσουμε τι γίνεται, πώ θα συντονιστούμε. Διότι θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι οι παράγοντε, όλοι αυτοί οι οποίοι ε, είναι αποδέκτες παραπώνων σε ε, κοινωτικό, σε ενωσιακό, σε εθνικό επίπεδο να δουν τι θα κάνουν αυτά τα προβλήματα κύριε ε, Πρόεδρε γιατί πριν από πολύ καιρό εγώ προείδρευα εδώ όπως εσείς στην Επιτροπή των Αναφορών και είχαμε τότε οργανώσει ε, μία συνάντηση με τον ε, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αλλά και τους Προέδρους των ε, Επιτροπών Αναφορών των Εθνικών Κοινοβουλίων και ακριβώς αυτό λέγαμε. Θέλαμε να αναζητήσουμε τρόπο του να επιλύσουμε το, το πρόβλημα τι θα πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει. Ε, γιατί είχαμε λάβει τότε κάποιες επιστολές. Τότε φτάσαν οι πρώτες. Για πρώτη φορά επομένως αυτό το σημερινό συζητούμενο πρόβλημα είναι απλά η συνέχεια γίνονται των συγκεκριμένων προβλημάτων τα οποία τα εγνωρίσαμε τότε πριν πολλά χρόνια. Διότι ο κόσμος πάει και χτυπάει στη λάθος πόρτα όταν αναζητούν άρρωγη βοήθεια, επανόρθωση των, των, όσων τους έχουν θυγεί. επομένω. αυτό θα πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο προσδοκούν, σε αυτό να κάνουμε κάτι. Και θα πρέπει επομένω. Ε, αν λάβουμε κάποια, κάποια τέτοια επιστολή διαμαρτυρία, θα πρέπει να την ε, ε, αναπέμψουμε εκεί που πρέπει, σε, νοσιακό ή σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό δεν είναι μονόδρομος. Όχι μόνο εμεί να στέλνουμε δηλαδή σε εθνικό επίπεδο. Και από το κάθε κράτος μέλο, από το, το εθνικό επίπεδο έρχονται σε εμά επιστολέ. αντίστοιχα. Άρα θα πρέπει να δούμε πρακτικά τι μπορεί να γίνει. Πώς θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τι νομικέ πτυχέ, τι θεσμικέ πτυχέ, ότι δεν μπορεί να κάνει από μόνο το πολίτη βέβαια και εμεί επομένω αυτό ασχίσουμε να δώσουμε μια απάντηση. Άρα, για να δούμε, για να δούμε σφαιρικά τι μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε να αναβαθμιστεί η συνεργασία μεταξύ διαμεσολαβητή, μεταξύ διαμεσολαβητή για του ανηλίκους, για τα θεσμικά όργανα που ασχολούνται με ανθρώπινα δικαιώματα και να δούμε επομένως πώς θα μπορέσουμε κάποια παράπονα, κάποιες καταγγελίες να τις ε, ε στείλουμε στους διάλογους που πρέπει και να δούμε με ποιες διαδικασίες θα γίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι για να δοθούν απαντήσεις θα πρέπει πρώτα κάποιος να καταλάβει πώς χειρίζονται τις καταγγελίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτοί που τις λάβουν, αυτοί που είναι αποδέκτες και να δούμε επομένως και ποιες πρακτικές συντρέχουν. Βεβαίω έχουμε εμπειρογνωμοσύνη εδώ, άφθονη. Και άρα θα μπορέσουμε να δώσουμε τι κατάλληλε και θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε πέρα του για τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων και σε εθνικό επίπεδο και σε ενωσιακό. Τώρα υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει να σα το τονίσω. Οι δικαστέ στα κράτη-μέλη. Ανέκαθαν, ήταν πάρα πολύ σημαντικοί είναι πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Άρα θα πρέπει να υπολογίζουμε και στη δική του βοήθεια όταν έρθει η ώρα τη υλοποίηση εφαρμογή του χάρτη, όποτε καλούνται οι δικαστέ να ερμηνεύσουν το κοινοτικό δίκαιο. Χέρι χέρι μαζί σα, κυρίε και κύριοι. Έχουμε εδώ σήμερα αυτούς του εκλεκτούς εμπειρογνώμονε για να τα συζητήσουμε. Και από ό,τι βλέπω ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και θα πρέπει βέβαια προσωπικά να ευχαριστήσω την πρόεδρο την κυρία Ματσόνη για το πόσο ενδιαφέρεται και, αλλά και είμαι σίγουρος, σίγουρη ότι και εσείς όλοι τα μέλη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής των Αναφορών ε, ενδιαφέρεστε πάρα πολύ γιατί είσαστε η κατεξοχήν ειδική ε, η Επιτροπή μάλλον η οποία περισσότερο από όλες ξέρει τι δεν πάει καλά σε αυτά τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η δική σας ε, συνεισφορά είναι πάρα πολύ σημαντική διότι έχουμε κοινή ευθύνη να δοθεί απάντηση στον πολίτη να δοθεί απάντηση σοβαρή διότι η απάντηση λυπάμαι δεν είμαι εγώ αρμόδιος για αυτό το οποίο ψάχνετε αυτό δεν αποτελεί απάντηση και μεγάλη μου χαρά βλέπω όλοι εδώ Ελπίζω όταν τελειώσει αυτή η συνάντηση να έχουμε σκεφτεί με ποιους τρόπους θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και έτσι οποιοδήποτε θεσμικό όργανο, οπουδήποτε θα μπορεί να δώσει την κατάλληλη απάντηση όταν λάβει μια καταγγελία ένα παράπονο και ο πολίτη θα πει ναι, ναι, κάποιος νοιάζεται για μένα. Επομένω, σα καλωσορίζω εσά και του ε, συνεργάτες οι οποίοι και βέβαια θα μου πούν πού κατέληξαν οι συζητήσεις μας. Ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο, την κυρία Ρέντι για την παρέμβασή της, γιατί υπογράμισε τα σημαντικά σημεία, τα πιο χρήσιμα, τα πιο σημαντικά ούτως ώστε όλοι μας να προβληματιστούμε και να βρούμε απαντήσεις μαζί. Όπως είπε η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ, είμαστε η εμπροστοφυλακή των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Είμαστε η Επιτροπή Αναφορών και το Γραφείο για τις καταγγελίες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγγελίες των πολιτών προ την Επιτροπή. Και το Κοινοβούλιο λοιπόν και η Κομισιόν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους πρέπει να απαντήσουν σε μια πλειάδα ανησυχιών των Ευρωπαίων πολιτών που εκφράζουν για τον τρόπο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. και η Επιτροπή Αναφορών και έχω το Γραφείο Καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τη συνθήκη. Έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα να συνομιλήσουμε τους πολίτες. Και οι πολίτες μέσω του εργαλείου αυτού της αναφοράς καταθέτουν τις αντιρρήσεις τους, τις αμφιβολίες τους, τις ανησυχίες τους, όχι μόνο προς το Κοινοβούλιο, αλλά προς όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών προβλέπει ότι το γραφείο της γραμματείας ξεκινάει μια διαδικασία και μια έρευνα που εμπλέκει όλα τα ενωσιακά όργανα. Έρχονται σε επαφή με τις εθνικές αρχές και τις τοπικές αρχές, κάνουν έρευνες επιτόπιες έρευνες και οι ευρωβουλευτές που είναι μέλη της Επιτροπής Αναφορών γνωρίζουν η σώμαση, ε, τι συμβαίνει, ποια είναι τα γεγονότα που καταγγέλλονται. Ο στόχος και η δραστηριότητα αυτής της Επιτροπής είναι να βρει ε, λύσει σε αυτά τα προβλήματα των ε, πολιτών. Λύσεις που δεν μπορούν από μόνοι τους οι πολίτες να βρουν όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Ρέντι, προσπαθούμε τουλάχιστον να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι αρμόδιος και να κατευθύνουμε τον πολίτη προς τον αρμόδιο. Το σημερινό σεμινάριο, το είπαμε και το επαναλαμβάνω, έγινε γιατί θέλουμε λίγο να ξεχερσώσουμε το πεδίο, ε, να δούμε πώς προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, ο χώρος αυτός μερικές φορές μοιάζει αρκετά συγκεχημένος. Δεν ξέρουμε μερικές φορές πότε όντως παραβιάζονται και πότε δεν παραβιάζονται οι... τα δικαιώματα των πολιτών. Εμείς λαμβάνουμε πάρα πολλές αναφορές και μας ζητούν την παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 56 ανοιχτές αναφορές. Και συχνά υπάρχουν ερμηνευτικές αμφιβολίες στις περισσότερες από αυτές. Όπως είπε και η κυρία Ρέντινγκ, ως πρόεδρος της Επιτροπής και εγώ, ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, συχνά στο παρελθόν οι πολίτες ζητούσαν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, απευθυνόμενοι προς την Επιτροπή Αναφορών ε, και προς άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Αυτά ήταν παλιότερα. Οι θεμελιώδες αρχές όπως εγγυώνται από την Χάρδα έχουν διαφορετικό ειδικό βάρος σήμερα. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε τα άρθρα της χάρτας μιλούν για τις θεμελιώδες αρχές από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην προστασία της ε, φυσικής ακαιρεότητα, της οικογένειας, της ιδιωτικής ζωής, των θεμελιωδών ελευθεριών, της ελευθερίας έκφρασης, ε, ενημέρωσης, πληροφορία, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το δικαίωμα πρόσβασης ε, στη δικαιοσύνη, της κυκλοφορίας, της κατοικίας. Είναι 54 τα άρθρα της χάρτας τα οποία ξεκαθαρίζουν με ξεκάθαρο τρόπο τις αρχές αυτές που αφορούν τον άνθρωπο. Και επειδή αναγνωρίζονται αυτές αρχές, ε, από την αναγνώρισή τους απορρέει και η προστασία. Αυτό όμως για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει μονοσήμαντη ερμηνεία. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη εγγύησης αυτών των ε, δικαιωμάτων. Δυστυχώς το πεδίο αυτό είναι αρκετά ε, χέρσο, αρκετά ε, συγκεχημένο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δίνουμε κατάλληλες απαντήσεις στους πολίτες. Το πρώτο σημείο είναι η ερμηνεία του άρθρου, του άρθρου 51 που προβλέπει, όπως είπε πολύ σωστά η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ, ότι οι διατάξεις της χάρτας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εργοποίηση του ενωσιακού δικαίου. Το επόμενο άρθρο, το 52, λέει ότι βασιζόμαστε την ε, σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και βασικών ελευθεριών. Αλλά όμως δεν εμποδίζει τίποτα και κανείς την Ένωση να ξεπεράσει το πλαίσιο της σύμβασης. Και σίγουρα αυτό περιπλέκει την, το καθήκον του ανθρώπου που ερμηνεύει τη χάρτα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνεργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γνωμοδοτήσουμε, να ενημερώσουμε. Πολύ συχνά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κοινοτική ευθύνη, κοινοτική αρμοδιότητα. Ε, συνέβη αυτό σε πάρα πολλέ αναφορές. Ε, μιλάμε για την ελευθερία τύπου, για την προστασία των ανηλίκων, για θέματα φύλου, ακόμα και για διακρίτηση λόγω ε, ράτσας. Εμείς προστατεύουμε πάνω απ' όλα το δικαίωμα της ηθαγένειας. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση βέβαια να δημιουργήσουμε προσδοκίες που δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε, αλλά και να δημιουργήσουμε και διαμάχες για θέματα αρμοδιότητας, που είναι πάρα πολύ δύσκολες να επιληθούν. Το βασικό είναι να δίνουμε μία μονοσήμαντη και χωρίς ε, αμφιβολίες ερμηνεία. Σήμερα μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και για να δώσουμε εγγύησεις ότι οι δράσεις μας θέτει πάντα στο κέντρο το συμφέρον του πολίτη. Γι' αυτό βασιζόμαστε στα κείμενα που έχουμε και κυρίως στη χάρτα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να ξεκινήσουν οι εργασίες του πάνελ μας. Θα σας παρουσιάσω την πρώτη ομιλήτρια. Πριν τους παρουσιάσω όμως, χαιρετώ την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ, η οποία αποχωρεί από τη συνεδρίασή μας. Την ευχαριστώ ακόμα μια φορά και την ίδια την Αντιπρόεδρο και την Κομισιόν εν το συνόλο της που θέλησε να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία της ε, Επιτροπής Αναφορών και του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, το πρώτο πάνελ. Τι σημαίνει στην πράξη ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Πώς θα μάθουν οι πολίτες, πότε εφαρμόζεται ο χάρτης. Αυτό είναι το πρώτο μας πάνελ. Χαιρετίζω εκ νέου τους ομιλητές που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση και που είναι εδώ σε αυτό το τραπέζι, η κυρία Μόνικα Φλασίκοβα Μπένοβα, ο καθηγητής Τζουζέπε Τεζάουρο, ο καθηγητής Σιέφ Φαν Ερπ, καθηγήτρια Έλσπεθ Γκίλτι και ο καθηγητής Ζων Πολζάκ Τους χαιρετίζω και θα δώσω καταρχάς το, ρόλο, το λόγο στην ε, κυρία Μπένουβα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει όλο και μεγαλύτερη σημασία στα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν θέλω υπερβολές, δεν μου αρέσουν, αλλά με ικανοποιεί πάρα πολύ να σκέφτομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση Θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι η συγγήτρια για την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου για την κατάσταση των Θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να σας απευθύνω το λόγο. Είναι πολύ διακεκριμένο το ακροατήριο. Η ατζέντα είναι σαφής, ο χάρτης ε, της, ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν ε, έχει νόημα να παραμείνει επί χάρτου. Πρέπει να αποκτήσει χρησιμότητα για τους πολίτες της Ένωσης και γι' αυτό πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη. Και για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή του, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν βασική γνώση του χάρτη και πότε ο χάρτης αυτός εφαρμόζεται. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό φαίνεται να είναι πρόβλημα. Γι' αυτό άλλωστε συναντηθήκαμε σήμερα. Σύμφωνα ε, με τα ευρήματα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, 72% των Ευρωπαίων πολιτών δεν αισθάνονται ότι είναι καλά ενημερωμένοι για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη. Θα πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή είναι ευθύνη, δική μας ευθύνη των ενωσιακών θεσμικών οργάνων για να είναι αποτελεσματικά τα δικαιώματα που αναφέρονται στο χάρτη, το, η κοινή γνώμη πρέπει να γνωρίζει ποια είναι και πώς τα προασπίζουν όταν παραβιάζονται. Καλύτερη διάβλη ε, επικοινωνίας, ε, πληροφορίας και δυνατότητας προσφυγής χρειάζονται. Καταρχήν τα δικαιώματα των παιδιών και των ε, ηλικιωμένων. Πολλές φορές δεν είναι γνωστό πώς θα προασπίσουν τα δικαιώματά τους, πού θα απευθυνθούν. Δεύτερον, και αυτό είναι γενικότερη παρατήρηση, υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με το τι, μπορεί, τι ρόλο παίζουν τα επιμέρους ένδικα μέσα. Η Κομισιόν αναφέρθηκε στις παρανοήσεις που υπάρχουν ε, και πολλές φορές ε, χαρακτήρισε τις περιπτώσεις αυτές ε, ως απόπειρες να χτυπήσουμε στη λάθος πόρτα. Χρειάζονται διευκρινήσεις. Όταν τα κράτη-μέλη ε, δρούν εκτός ευρωπαϊκής... Τα κράτη-μέλη έχουν και την εθνική νομοθεσία και εάν οι πολίτες θεωρούν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί πρέπει να είναι βέβαιοι ότι η προσφυγή τους γρήγορα θα φτάσει τα αρμόδια ε, τοπικά δικαστήρια ή τους οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσφέρει ένα άλλο επίπεδο προστασίας αφού έχουν εξαντληθεί τα εθνικά ένδικα μέσα. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Κομισιόν δεν είναι δικαστήριο, δεν είναι εφετείο κατά των αποφάσεων που λαμβάνουν τα εθνικά ή διεθνή δικαστήρια, εκτός από την ενημέρωση για το χάρτη, άτομα που θεωρούν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πρακτική πληροφόρηση για τα ένδικα μέσα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προωθήσουμε τα εργαλεία που υπάρχουν, τα μέσα που υπάρχουν, ενημερώνοντας την κοινή γνώμη για το ποιος είναι ο αρμόδιος ε, ανάλογα με την προσφυγή. Το e-Justice Portal της Ευρώπης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πρέπει όμως να προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες ε, και τις δυνατότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Το Portal θα πρέπει να δίνει πληροφορίες στην κοινή γνώμη για τα ένδικα μέσα σε περιπτώσεις ε, παραβιάσεων ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης το πόρταλ θα πρέπει να λειτουργεί μια πλατφόρμα ενημέρωσης σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στην περίπτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να το κάνει αυτό από κοινού με το με την Ευρωπαϊκή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, τα, τους οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο, ε, και βεβαίως με βάση την ομολογία των δικαστηρίων, των αρμοδίων δικαστηρίων και μαζί με άλλα, ε, άλλους φορείς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, αν δεν εφαρμόζεται ο χάρτης, η Κομισιόν εξηγεί πως η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα κράτη-μέλη μπορεί να, ε, να διοχετευθεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Είναι ρόλος μας ε, σε αυτό το σεμινάριο σήμερα να δούμε πώς θα θεσπίσουμε ε, και θα κάνουμε θεσμικό ένα τέτοιο μηχανισμό. Διάφορα σημαντικά βήματα έκανε η Κομισιόν που ενημέρωσε την κοινή γνώμη για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών. Κάποια πράγματα πρέπει να αναφέρουμε εδώ. Ε, έχει ε, κάνει περισσότερες δραστηριότητες σε σχέση με τον ρόλο της Ένωσης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις δυνατότητες παρέμβασης που υπάρχουν. Η Κομισιόν θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι διατίθενται ε, εξηγήσει στους προσφεύγοντες και στα ενδιαφερόμενα μέρη ανάλογα με τις ανάγκες. Μίλησα ήδη, ήδη για τα δικαιώματα των παιδιών που συχνά δεν είναι πολύ γνωστά. Έτσι θα ήταν ευκταίο να υπάρξουν γραπτός επεξηγήσεις με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά. Ε, η Κομισιόν ε, περιλαμβάνει και ένα ε, θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα παράρτημα με συχνά, ε, συχνές ερωτήσεις. Επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση των δικαστικών και άλλων νομικών αρχών. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε αστικά και εμπορικά θέματα και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για ποινικά θέματα και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Δικαιοσύνης. Συμπεραίνοντας θα ήθελα να κάνω μια βασική παρατήρηση που αφορά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Η πρόσφατη κρίση στην Ευρωζώνη σίγουρα δημιουργεί τάσεις από σύνθεση της Ένωσης. Όλο το ευρωπαϊκό εγχείρημα φαίνεται να απειλείται. Έτσι νομίζω. Σίγουρα ρόλος μας είναι να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσεγγίσει όσο γίνεται περισσότερο τους πολίτες. Ένας τρόπος ε, είναι μπροστά μας, μπορούμε να ενημερώσουμε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την, ε, τους αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας τους. Δεν είναι δυνατόν να ε, επεξεργάζονται μόνο το 1 τρίτο των προσφυγών. θα πρέπει να εξηγηθεί η εφαρμογή του χάρτη Ε, είναι πολύ δυσάρεστο να μην προχωρούμε γρήγορα σε αυτούς τους τομείς, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τόσα καθήκοντα και προκλήσεις για να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ότι θα είναι αποτελεσματικές οι συζητήσεις στο σεμινάριο. Εύχομαι επικοδομητικές, γόνιμες συζητήσεις και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας κυρίες και κύριοι. Ε, και εγώ σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να ενημερώσω όλους σας ότι καταρχάς θα μιλήσουν πρώτα όλοι οι προσκεκλημένοι μας και εν συνεχεία θα δώσουμε τη δυνατότητα για ερωτήσεις ε, από τους ε, ευρωβουλευτές. Αλλά και οι εμπειρογνώμενες μπορούν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Θα έχουμε λοιπόν έχουμε στη διάθεσή μας συνολικά 45 λεπτά για αυτό το θέμα. Ο μισός χρόνος είναι για τους ομιλητές μας και ο μισός για ερωτήσεις. Ο κύριος Τεζάουρο, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτή την προσπάθεια κοινού προβληματισμού. Είχα την τιμή Στα 30 χρόνια να ασχοληθώ με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο ΔΕΚ τότε και σήμερα στο Ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως όλα τα νομικά κείμενα, είναι απλώς ένας χάρτης. Θα πρέπει να αποκτήσει ζωή κάθε μέρα από τους νομικούς, από τους δικαστές, αλλά όχι μόνο από αυτούς, και από τους νομοθέτες, από τους διοικητικούς υπαλλήλους, από όλους όσους συνεισφέρουν προκειμένου να αποκτήσει σάκα και οστά αυτό το σημαντικό εργαλείο. Ο χάρτης δημιουργήθηκε μετά από, μια μεγάλη, μετά από μια μεγάλη προσπάθεια και μια μακρά περίοδο όπου το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων προέκυπτε πιο ανάγλυφα από την ομολογία. Διότι ξέρετε ότι οι συνθήκε δεν έλεγαν τίποτα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο χάρτης δεν προέκυψε ξαφνικά μία νυχτή. Έζησε σε ένα λίμπο που δημιουργήθηκε από μία παράδοξη συνένεση, έζησε για μία δεκαετία σε μία κατάσταση έτσι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι. Στην πραγματικότητα ήταν μια Γάλλη όμω ερμηνευτική παρηγοριά. Δεν θέλω να πω πνευματική. Πολύ σημαντική λοιπόν. Για όλους όσους ασχολούνται με τον κλάδο του κοινοτικού δικαίου. Με την ε, Λισαβόνα έγινε ένα εργαλείο και νομικά δεσμευτικό πια. Τι καθόρισε η Λισαβόνα. Ε, λειτουργήσε όπως ε, το άνοιγμα μιας, ε, ενός μπουκαλιού σαμπάνιας. Δηλαδή, οι προσδοκίες ήταν πάρα πολλές. Γιατί πολλοί λέγανε ο χάρτης δεν είναι τίποτα, δεν έχει αξία, αλλά αυτό δεν ήταν αλήθεια. Με τη Λισαβόνα προέκυψε κάτι παραπάνω αλλά δημιουργούν και πολύ περισσότερες προσδοκίες από αυτό που ήταν ε, στο χάρτη. Συχνά ο τύπος, αλλά όχι μόνο ο τύπος, δημιουργεί προσδοκίες. Και όταν αυτές οι προσδοκίες δεν υλοποιούνται, φυσικά υπάρχει μια στιγμή που αισθανόμαστε κενοί, ένα άδειασμα. Αυτή είναι η σημερινή στιγμή, όπου όλοι θεωρούσαμε ότι επειδή ήμασταν ε, κακοπληροφορημένοι, ότι η συνθήκη της νίκαιας θα αποτελούσε ένα απόλυτο εργαλείο, ο χάρτης μάλλον της νίκαιας, θα ήταν ε, ένα μέσο απόλυτης προστασίας. Υπήρχε ένα πρόβλημα εφαρμογής του χάρτη της νίκαιας, ε, που που είναι το ίδιο με το θέμα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, γιατί δεν εφαρμόζεται πάντα. Το κοινοτικό δίκαιο δεν θέλουμε πάντα, δεν θέλουν πάντα όλοι να εφαρμοστεί. Στο χάρτη, όπως και στα δύο κείμενα που προέκυψαν από τη μεταρρύθμιση με τη Λισαβόνα, υπενθυμίζουμε τρόπο σχεδόν μονομανή την έλλειψη καινοτομία του χάρτη σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ιδίως ό,τι αφορά τις ε, αρμοδιότητες που έχει επ' αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πώς θα τα εξηγήσουμε στον πολίτη. Όταν μη, μη διηγηθήκαμε το παραμύθι ότι ο χάρτης το, της νίκιας θα ήταν η πανάκια για όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πώς θα μπορούμε να εξηγήσουμε στον πολίτη όπου ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ο χάρτης της νίκης γιατί απλούστατα δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο. Φανταστείτε μία περίπτωση ότι μερικές φορές εκεί που υπάρχει κοινοτικό δίκαιο ισχύει και ο χάρτης της νίκης, ισχύει, ισχύει και το κοινοτικό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο. Πολυεπίπεδη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και πήγαινε να εξηγήσει ότι όποιο εργαλείο δίνει τη μεγαλύτερη προστασία, εκείνο είναι αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν αρκούν δέκα λεπτά για να εξηγούμε κάθε φορά, να εξηγήσουμε τους λόγους αυτής της μεγάλης αυταπάτης. Η μεγάλη αυταπάτη οφείλεται στον τύπο. Γιατί ο τύπος δεν θέλει ημίμετρα. Θέλει κάτι το συγκλονιστικό. Θέλει νέα χτυπητά, βαρβάτα. Το γεγονός ότι ο χάρτης της νίκης έγινε συνθήκη, αλλά εφαρμόζεται όμως μόνο στο βαθμό που εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο, αυτό δεν είναι μεγάλο νέο, είναι κάτι φυσιολογικό, καθημερινό. Και οι ειδήσει ε, των εφημερίδων ε, και οι εφημερίδες γενικά ζουν από τα ασυνήθιστα. Οι καθηγητές που μιλάνε στους φοιτητέ έχουν επίσης μεγάλη ευθύνη, μιλάνε στους νέους και λένε στους νέους ποιος είναι, ποια είναι η οδός για να εφαρμοστεί ο χάρτης της νίκης για να φτάσουμε σε μια πραγματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι καθηγητές εφήβραν τα ε, το κοινοτικό δίκαιο. Ορισμένοι δεν ξέρουν καν περί τίνος πρόκειται και πηγαίνουν απλώς και συμμετέχουν σε συζητήσεις, σε συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, στα, στα πανεπιστήμια κτλ. Μιλάνε για αυτό που θα θέλανε οι ίδιοι. Δεν μιλάνε για την πραγματικότητα. Είναι μεγάλη ευθύνη των εκπαιδευτικών, των καθηγητών. Γιατί αυτή η μετάδοση της γνώσης στους νέους είναι μια τεράστια ευθύνη. Γιατί οι νέοι τα απορροφούν όλα αυτά. Απορροφούν όλα όσα τους διηγούνται. Ο τρόπος που διαδίδονται τα νέα είναι πάρα πολύ γρήγορα. Οι δικαστές και οι δικηγόροι και όλοι θεωρούσαν ότι ο χάρτης της νίκαιας ήταν το απόλυτο εργαλείο για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι πρώτες αποφάσεις, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και αλλού, αρκεί να διαβάσετε την ομολογία του ΔΕΚ σας δίνει να καταλάβετε ότι αυτός ο, αυτή η τάση τελικά διαμορφώνονταν σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, ο χάρτης της νίκαιας πέρα από την άμεση εφαρμογή δημιουργεί και μια μεγάλη διαλεκτική για τη διαφορά μεταξύ ε, θεμελιωδών αρχών, ε, κλασικών κανόνων, μια σειρά από... Αυτές είναι, μια, είναι μια σειρά από περιττές συζητήσεις. Γιατί αρχίζαμε να προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το χάρτη τη νίκη εκεί όπου δεν έπρεπε να εφαρμοστεί. Έχω, υπάρχει λοιπόν η τεράστια ευθύνη των δικαστών και των δικηγόρων. Ειδικά σε εμά στην Ιταλία, για διάφορου μήνε είχαμε μια διαφορά μεταξύ των κλασικών ε, δικαστών και του συνταγματικού δικαστηρίου. Διότι το συνταγματικό δικαστήριο τους ε, προειδοποίησε από την αρχή. Προσοχή, πάτε πολύ μακριά στην εφαρμογή του χάρτη τη νίκη. Και τώρα ηρεμήσαμε κάπως. Πέσανε οι τόνοι. Δεν υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός ό,τι αφορά την εφαρμογή του χάρτη της νίκαιας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Εγώ θα ξεκινούσα από την τελευταία παρατήρηση της κυρίας Μπένοβα. Κατ, κατ' εμένα πρέπει να ξεκινήσουμε να μιλάμε από τα μικρά παιδιά. Θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε εγχειρίδια με με ανθρωπάκια να εξηγήσουμε τι είναι το ναι. κοινοτικό δίκαιο, τι είναι ο χάρτης της νίκης και πώς είναι, είναι σημαντικό να ζούμε μαζί. Άντρες και γυναίκες διαφορετικής προέλευσης, διαφορετικής κουλτούρας. Εν συνεχεία θα πρέπει να πάμε στους επαγγελματίες, δικηγόρους και δικαστές. Για, οι, δικαστές γενικά έχουν ένα τεράστιο πλαίσιο μέσα στο οποίο καταρτίζονται κτλ. Αλλά όχι οι δικηγόροι. Αλλά οι δικηγόροι είναι το interface ανάμεσα στην, ε, στο κοινοτικό επίπεδο και στους πολίτες. Πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ στην κατάρτιση των δημοσιογράφων, των δικηγόρων και των δικαστών. Γιατί ο βαθμός γνώσης... Τέλος Αφήστε τους καθηγητές, εγώ είμαι καθηγητής και δεν θέλω να μιλήσω για αυτούς. Αλλά για τους επαγγελματίες του δικαίου, που είναι το φίλτρο μεταξύ των πολιτών και των εργαλείων προστασίας των δικαιωμάτων, ε, αυτούς πρέπει να τους ε, καταρτήσουμε. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε σε πόρους, σε χρόνο, σε, σε προσπάθεια, ειδικά εκεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Τεζάουρο. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή νομική κουλτούρα ε, των επαγγελματιών του δικαίου και χθες εγκρίθηκε ένα πιλωτικό σχέδιο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για την κατάρτιση ακριβώς των επαγγελματιών. Ε, προσυπέγραψα και εγώ. Πηγαίνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαι πολύ ικανοποιημένη λοιπόν που συμφωνούμε με τις ανα... ως προς τις ανάγκες τουλάχιστον. Τώρα πάμε στον καθηγητή Σιεφ Φανέρπ από το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ. First Πρώτα πρώτα, να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας, κυρίες και κύριοι. Όταν συζητούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνήθω, μιλούμε για τον ιδιωτικό βίο, τους ανηλίκους, όμως είναι και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα που είναι τόσο άσχημη οικονομική συγκυρία. Και είδατε ότι η τράπεζα τράπεζα στο κιλό του γκρεμού. Σοβεί αυτή η τραπεζική χρήση. που θα πρέπει να δούμε τι ποια είναι τα δικαιώματα των πολιτών εν, εν μέση κρίση. Σε σχέση λοιπόν πάντα με την ε, ιδιοκτησία. Και έχουμε το άρθρο 17 του χάρτη που ορίζει, περιγράφει το γεγονός στην ιδιοκτησία και ορίζει ότι όλοι έχουν το δικαίωμα εις το να κατέχουν, διαθέτουν ε, όπως θεωρούν ε, ότι τους ανήκει νομίμως. Επομένως, θα πρέπει να ληφθεί βέβαια το υπόψη το δημόσιο συμφέρον και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, κάθε φορά το τι άλλη διάταξη δικαίου υπερισχύει. βεβαίω και αυτή η διάταξη στηρίζεται στο, στη Σύμβαση των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων στο σχετικό άρθρο και επίσης έχουμε και το άρθρο 70 ή 17 που λέει ότι εξαρτάται το τι θα ρυθμιστεί και από την ομολογία. Να, για να δούμε επομένω τι ορίζει το κοινοτικό δίκαιο, διότι είπαμε ότι ο χάρτης ε, ισχύει ε, πάντα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό έγινε πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και την απόφαση Χάουαρτ του 1979. Τότε όρισε το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι πρόκειται για δικαίωμα το δικαίωμα τη ιδιοκτησία ή στα πλαίσια του κοινωτικού δικαίου. Και επίση θα ήθελα να σα τονίσω ότι ήδη έχουμε διατάξει του κοινωτικού δικαίου που ορίζουν σχετικά. Ε, κυρίως έχουμε οικονομικό δίκαιο όπως ακριβώς ε, ε, ο κανονισμός για την πτώχευση όμως πέραν αυτών όλων έχουμε έχουμε τώρα το 345 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι το, το, το, το, δικαίωμα στην κυριότητα είναι δικαίωμα είναι, είναι θέμα που ρυθμίζεται στο εθνικό δίκαιο οπότε αυτό παρά αυτή την ευρεία διατύπωση τελικά όλα αυτά σημαίνουν ότι η εθνικοποίηση, η ιδιωτικοποίηση, όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα των κρατών μελών. Βέβαια θα πρέπει να δούμε ε, όλα αυτά ε, πώς επιδρούν επί του Ευρωπαίου. Είπαμε ότι έχουμε τις οδηγίες, έχουμε τους κανονισμούς, ε, έχουμε τον κανονισμό για την επτόχευση. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το πράγματο δίκαιο. Όμως, όμως είναι δυνατόν να θυγούν τα δικαιώματα και με άλλο τρόπο τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων. Να σας πω, τι να σας πω τώρα, έχω 10 λεφτά και θα απλώς να σας υποδείξω δύο προβληματάκια μπορεί να ανακύψουν πρώτα-πρώτα. έχουμε τις τέσσερις ελευθερίες της εγκατάστασης, ε, ας πούμε η ελευθερία του κανείς να μπορεί να αγοράσει μια δεύτερη κατοικία εκτός της χώρας στην οποία διαμένει. Και έχουμε εδώ πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και να σας πω ένα παράδειγμα ε, όπου έχουμε κάποιον αγοραστή δεύτερης ε, κατοικίας ή στην Ισπανία τα αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα εκεί στην, ε, στην παραλία γιατί εκεί πέρα υπάρχει μια διάταξη δημοσίου δικαίου όσον αφορά την κυριότητα και δεν εγνώριζαν ότι υπάρχει αυτός ο περιορισμός οπότε το αποτέλεσμα ήταν στο ότι ε, τους απολωτριώθηκαν οι κατοικίες που αγόρασαν και χωρίς να λάβουν την δέουσα αποζημίωση. Οπότε αυτό ε, είναι πρόβλημα για τους αλλοδαπούς που να αγοράσουν σπίτι, αλλά το πρόβλημα είναι για τους Ισπανούς που θέλουν να διαθέσουν ένα κίνητο. Πάντως όταν αφορά κάποιον αλλοδαπό τότε είναι θέμα κοινωτικού δικαίου και τότε ακριβώ μπαίνει στο παιχνίδι και ο χάρτης. Επομένως θα έπρεπε να ληφθεί πρωτοβουλία από πλευρά Ευρώπη και έτσι όλοι αυτοί οι περιορισμοί να είναι γνωστότεροι ούτω ώστε να είναι γνωστά ε, το, το τι πρόβλημα να προκύψουν σε σχέση με το δικαίωμα ή στην κυριότητα του άρθρου 17. Και αυτό αφορά όμω και ε, τα ευρωπαϊκά δεσμικά όργανα που θα πρέπει ακριβώ και αυτά να αποφύγουν το να παραβιάζουν αυτό το δικαίωμα και θα πρέπει να φροντίσουν το πώ θα υπάρχει περισσότερη διαφάνεια για αυτέ τι δημοσίου δικαίου χαρακτήρα διατάξει. Υπάρχει τώρα και άλλο ένα πρόβλημα και, άλλο, και άλλο θέμα ε, που αφορά τι συντάξει το δικαίωμα στην συνταξιοδότηση. Διότι υπάρχει πίεση λόγω τη ε, οικονομική κρίση. Πιέζονται οι κυβερνήσει, πιέζονται τα συνδικάτα, πιέζονται οι οργανώσει των συνταξιούχων να δεχθούν την περικοπή των συντάξεων. Τώρα, η σχετική νομολογία είναι σαφής. Ότι όταν υπάρχει προσδοκία, η προσδοκία, η απλή, δεν προστατεύεται. Όμως, κανείς έχει πληρώσει κάποιες εισφορές. Εκτός τα λεφτά του και επομένως θα πρέπει να δικαιούται σε σύνταξη. Όμως, σε αυτή την κατάσταση οικονομική της πραγίας ίσως δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά η περικοπή των συντάξεων αυτό όμως θα πρέπει να είναι το τελευταίο καταφύγιο, τελευταία λύση. Εδώ λοιπόν τι ρόλο παίζει ο χάρτης. Οι Υπουργοί Οικονομικών κάθονται και συζητούν τα μέτρα της λιτότητας Δεν μπορείς να πει ότι θα πρέπει του κάθε κατωσμένου κάτι να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 και η βλάβη αποκαταστάθηκε και συνεχίζουμε. Για να συνοψίσω, λέει ο μιλητή, τι είπα προηγουμένω πριν συνεχίσω παρακάτω. Σας ανέφερα την περίπτωση των δικαιωμάτων των στεξιωτικών. Βεβαίω και είναι δικαίωμα ενός κράτους να έχει ένα συνεξιωτικό σύστημα το οποίο είναι συγκροτημένο όπως θεωρείται καλύτερα. Και αυτό ισχύει επίσης και για τις κοινωνικές παροχέ, Επιδόματα κλπ. Ο άπαξ όμως και το σύστημα αυτό ισχύει και υπάρχουν οι εισφορές και υπάρχει η προσδοκία τότε είναι γεγονός αυτό το δικαίωμα και έχει οικονομικό περιεχόμενο. Οπότε, αυτό αποτελεί αντικείμενο κυριότητος την ταινία του άρθρου 17 και του υπαριθμών 1 της ε, σύμβασης. Αυτή λοιπόν η ιδιοκτησία του δεν είναι δυνατόν να τους αφαιρεθεί. Τώρα όμως, όταν η οικονομία σου δώσει καλή κατάσταση, δεν υπάρχει εναλλακτική. Όμως είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι η τελευταία λύση, η τελευταία, το τελευταίο βήμα. Έχουν δικαιώματα όμω και σε περίπτωση κατάρρευση της οικονομίας οι πολίτες. Ακριβώς και τότε. Και ιδίω εκείνοι οι οποίοι είναι είναι ηλικιωμένοι και έχουν δικαίωμα σε σύνταξη. Είναι εκείνοι οι οποίοι δούλεψαν για αυτές τις συντάξεις, έχτισαν αυτή την ε, κοινωνία στην οποία ζούμε. Βεβαίω έχουμε και το άρθρο 25, το οποίο λέει σε σχέση με τα δικαιώματα των ηλικιωμένων ότι αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σέβεται το δικαίωμα των ε, ηλικιωμένων να ζουν μια ζωή αξιοπρεπή, ανεξάρτητη και να μπορούν να συμμετάσχουν στι διαφορετικέ πτυχέ τη ζωή. Πώ όμω κανεί να είναι έτσι ανεξάρτητο, εάν οι συντάξει οι οποίε ε, έπρεπε να καταβληθούν αφαιρούνται. Αυτό βέβαια είναι ακροβασία. Ακροβασία σε λεπτό σκηνή και ε, θα πρέπει να το προσέξουμε. Και ακριβώ όπως είπα πριν την ε, βλάβη του χειρικού συστήματος, να δούμε πού υπήρχε το ρόλο τη Ευρώπη. Όταν έρχονται οι Υπουργοί Οικονομικών και απαιτούν από τα κράτη-μέλη να λάβουν κάποια μέτρα λιτότητα, το ότι υπάρχει παρέμβαση ε, και ακριβώ σε αυτό το σημείο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίω ε, εσεί που εκπροσωπείτε τους πολίτες θα πρέπει να φροντίσετε εκείνοι οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι και πολλές φορές δεν ακούει τη φωνή τους ότι αυτοί θα την χάνουν τις προστασίες Σας ευχαριστώ. εγώ σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ζητώ συγγνώμη για το πρόβλημα που είχαμε τα μικρόφωνα. Η κυρία Έσπελ τώρα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να σας μιλήσω σήμερα για ένα τεραστίο ενδιαφέροντος θέμα. Δηλαδή πώς θα κάνουμε γνωστό το χάρτη και θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν να λυθούν με το χάρτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα αρχίσω με ένα παράδειγμα, όπως λέει και το πρόγραμμα. Μια, ένα βράδυ με έβγαλαν έξω, με χτύπησαν, δεν ξέρω γιατί. Μας πήγαν σε ένα χώρο όπου ήταν τηλέφωνα σε μια μικρή αίθουσα, μας χτύπησαν, μετά ήταν δύο, μετά ήρθαν και άλλοι δύο. Αυτό έγινε τη νύχτα. Είμαστε 4-5 που δεν κοιμόμαστε, κάναμε θόρυβο, φωνάζαμε, γιατί είχε τρελαθεί ο κόσμος και είμαστε σε άσχημη κατάσταση. Μας έβγαλαν έξω γι' αυτό. Αυτό έγινε πριν από μια εβδομάδα. Ήταν πολλοί, με χτύπησαν με ε, ραβδί, με κλόμπ, ε, τρεις-τέσσερις ε, αστυνομικοί, με χτύπησαν στο μυρό δύο-τρεις φορές. Πρόκειται για τη Λιβύη του Καντάφη, δυστυχώς όχι. Είναι λυπηρό αυτό είναι μια προσφυγή από ένα συνόδευτο παιδί το οποίο το στην Ελλάδα. Ε, αυτή είναι αναφορά του παρατηρητήου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκδόθηκε 31 30 Σεπτεμβρίου φέτος. Αυτός ο ισχυρισμός ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την έκθεση του Έλληνα διαμεσολαβητή για τις συνθήκες κράτησης αλλοδαπών στην Ελλάδα Υπάρχουν και τρεις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα. Υπάρχουν και από τον ε, ε, από την Επιτροπή κατά των βασανιστήριων αναφορές ε, από τον συνήγορο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, τι αναφερόταν ε, στην έκθεση αυτή. Η Frontex, η οποία ελέγχει και συντονίζει τα, τους συνοριοφύλακες ε, για να ελέγξει την παράνομη είσοδο ε, μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα, γνωρίζει ότι όσοι παραδίδονται ε, θα τεθούν υποκράτηση σε συνθήκες που παραβιάζουν το άρθρο 4 του χάρτη, δηλαδή την απαγόρευση βασανιστήριων ή ε, τιμωρίων ή αναξιοπρεπούς ε, συμπεριφοράς. Αυτό τώρα ε, καλύπτεται από το χάρτη. Στην απάντηση σε έναν ανακοινωθέν τύπου το Σεπτέμβριο από τη Frontex ήταν ότι αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, ότι οι συνθήκες κράτησης στα ελληνικά κέντρα κράτηση αλλοδαπών είναι θέμα εθνικής νομοθεσίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις εθνικές αρχές. Γι' αυτό λοιπόν το άρθρο 4 του χάρτη δεν εφαρμόζεται. Και η απάντηση της Frontex είναι ότι δεν θεωρεί ότι πρέπει να δώσει οδηγίες στους συνοριοφύλακες των κρατών μελών που εργάζονται υπό την Frontex τα ελληνοτουρκικά ε, σύνορα θα πρέπει να σταματήσουν να παραδίδουν τους κρατούμενους στους Έλληνες ε, αξιωματικούς. Η Επίτροπος Μάλστρομ επίσης εξέδωσε δήλωση στο blog της στις 22 Σεπτεμβρίου απαντώντας την έκθεση αυτή και επιβεβαιώνοντας ότι είχε κάνει συζητήσεις με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το θέμα αυτό και ότι θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στην Ελλάδα ώστε η τελευταία να βελτιώσει τις συνθήκες κράτησης στο έδαφος της. Ε, συμφωνεί όμως με την Frontex και εκείνη ότι το θέμα αφορά την ε, εθνική νομοθεσία. Ο Γενικό Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε μια απόφαση που ονομάζεται ΕΝΕΣ ε, γνωμοδότησε, δεν έχει υπάρξει απόφαση του δικαστηρίου ακόμα, σχετικά με το αν ένας ετών άσυλο, ο οποίος ε, ε, προσφεύγει κατά της βρετανικής απόφασης με βάση τον Dublin 2 να τον γυρίσει στην Ελλάδα, αν η προσφυγή του καλύπτεται από την κοινοτική νομοθεσία. Ο Γενικός Εισαγγελέας Τρασένιακ θεωρεί ότι πράγματι ο χάρτης εδώ εφαρμόζεται και ειδικότερα το άρθρο 4 στο φως των συνθήκων κράτησης ε, που έχουν καλά τεκμηριωθεί ε, και αφορούν την Ελλάδα. Πρέπει να, έχει, να υπερέχει ο χάρτης σε σχέση με τις ρυθμίσεις του Δουβλίνου και ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να στέλνουν ετούντες άσυλο από ένα κράτος μέλος ένα όπου είναι αξιοπρεπείς οι συνθήκες υποδοχής σε ε, ένα άλλο κράτος μέλος στην Ελλάδα προκειμένου και που έχει συνθήκες κράτησης που παραβιάζουν το χάρτη. Έτσι λοιπόν η, αυτή είναι η γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε εάν και το δικαστήριο θα συμφωνήσει μαζί του. Πάντως ο Εισαγγελέας θεωρεί ότι οι συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του χάρτη όταν μπαίνει το θέμα του πού θα πρέπει να υποβάλουν τις ε, προσφυγές τους οι αιτούντες άσυλο και τη συνέχεια θα δοθεί σε αυτές. Είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε από την έκθεση του παρατηρίου του για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι ε, οι Γερμανοί συνοριοφύλακες που συμμετείχαν στη δράση στα, στη ελληνοτουρκικά σύνορα, όταν αυτοί λοιπόν συνειδητοποίησαν τις συνθήκες κράτησης, ζήτησαν από τους ανωτέρους τους στο Βερολίνο να τους εξουσιοδοτήσουν να μην παραδίδουν κρατουμένους που περνούν τα σύνορα στις ελληνικές αρχές. Κατά συνέπεια, οι Γερμανοί συνοριοφύλακες που μετήχαν σε αυτή την επιχείρηση δεν εργάζονται, δεν αναλαμβάνουν εκεί αυτά τα καθήκοντα. Ε, αυτοί οι πολίτες της Ένωσης θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να καλούνται να παραβιάζουν το άρθρο 4 του χάρτη. Από του παρόντος όμως, τι ένδικα μέσα υπάρχουν. Η απάντηση που δίνουν τα θεσμικά όργανα είναι μια απάντηση που δεν ικανοποιεί. Η Frontex θεωρεί ότι είναι θέμα εθνικού δικαίου αυτό θα δίνουμε οδηγίε στους συνοριοφύλακες ε, που εργάζονται σε επιχειρήσει στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας να παραδίδουν ε, τους κρατουμένους κράτηση τους πρόσφυγες αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τη θέση αυτή. Στις 7 Σεπτεμβρίου φέτος ε, το PDC αποκάλυψε ότι σε απάντηση μιας αδημοσίευσης έκθεσης ακόμα από τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των κρατουμένων στο Αφγανιστάν, ο επικεφαλής Νέιζο, επικεφαλής των, του στρατού των δυνάμεών μας στο Αφγανιστάν, απαγόρευσε την παράδοση των κρατουμένων από το, το, τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στις αφγανικές αρχές λόγω των συνθήκων ε, που επικρατούν εκεί. Πάλι εδώ πρόκειται για θέμα που αφορά το άρθρο 4 του χάρτη. Δεν μπορείς να παραδίδεις ανθρώπους σε άλλες αρχές γνωρίζοντας ε, ή έχοντας βάσιμους λόγους να υποθέτεις ότι θα υποστούν ε, βασανιστήρια ή θα τιμωρηθούν ή θα αντιμετωπιστούν με τρόπο αναξιοπρεπή. Ε, έτσι λοιπόν τώρα έχουμε μια μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το άρθρο 4 του χάρτη το οποίο εφαρμόζεται και την χάνει σεβασμού από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν ε, αφού δεν μπορούν να παραδίδουν κρατουμένους και αυτοί είναι άνθρωποι, αντίπαλοι τους που τους πυροβολούν οι Αφγανοί τους ε, ανθρώπους του ΝΑΤΟ. Ενώ έχουμε συνοριοφύλακες στον Εύρο που συντονίζονται από τη Frontex και ισχυρίζονται ότι δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4. Αυτό υποδηλώνει υπακριβώς πόσο σκληρά πρέπει να δουλέψουμε αν θέλουμε να εφαρμόζεται αποτελεσματικά, ε, αποδοτικά ο χάρτης και να προστατεύει και τα συνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα, όπως και τους ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν ένα δεύτερο σπίτι σε άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συνεχίσουμε αυτό που έλεγαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Θέλω να πω πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα ε, για να σας δείξω ότι σε αυτή την ελληνική υπόθεση το Βέλγιο καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Στρασβούργου γιατί εφάρμοσε τον κανονισμό του Δουβλίνου και απέστειλε στην Ελλάδα άτομα τα οποία είχαν εισέλθει παράνομα από την Ελλάδα και φτάσαν στο Βέλγιο. Είμαστε σε μια περίπλοκη λοιπόν κατάσταση. Καταρχάς αυτό είναι παράδοξο, γιατί ο χάρτης δημιουργήθηκε ως ένα εργαλείο το οποίο θα απλούστευε τη ζωή των πολιτών. Πριν το χάρτη, τα θεμελιώδη δικαιώματα εγγυόνταν βάσει μιας ε, πολύ περίπλοκης νομολογίας του 10 που οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν ήξεραν, ήξεραν μόνο οι εμπειρογνώμονες, μόνο οι ειδικοί. Γι' αυτό ακριβώς θέλαμε μια δήλωση, μια διακήρυξη, κάτι το σαφές και θυμάμαι ότι η σύμβαση μέσω του Βρετανού τότε εκπροσώπου έλεγε ότι θα πρέπει να μπορούμε να βάζουμε αυτό το χάρτη σε, όλες, όλα τα αστυνομικά τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο ώστε όλοι οι πολίτε να γνωρίζουν τα δικαιώματά του. Κι όμω, ο χάρτη επαύξησε την, ε, το πρόβλημα και την περιπλοκότητα του τοπίου αυτού. Να σας δείξω πόσο περίπλοκο είναι αυτό ε, με δύο παραδείγματα. Καταρχάς έχουμε πάρα πολλές πηγές ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το άρθρο 6 στη συνθήκη αναφέρει το χάρτη. Υπάρχουν οι γενικέ αρχές του δικαίου επίση, τις διατηρήσαμε, που είναι οι κοινέ ε, συνταγματικές συνθήκες, από τις κοινέ συνταγματικές συνθήκες μέχρι τη σύμβαση. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως εφαρμόζεται μέσω τη χάρτας, που τα εγγυώματά τη τα εγγυάται η σύμβαση. Και εν συνεχεία μετά την ε, προσφυγή που θα υπάρχει η Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς μπορείτε να περιμένετε ο δυστυχή πολίτης να καταλάβει ποια είναι τα δικαιώματά του μέσα από αυτή την, τον πολλαπλασιασμό των κειμένων. Και το δεύτερο πρόβλημα που το αναφέραμε, αλλά είναι ακόμη πιο περιπλοκό από ό,τι αναφέρουμε, είναι σε τι εφαρμόζεται ο χάρτης. Εφαρμόζεται στους, ε, στα θεσμικά όργανα της ε, Ένωσης, αυτό είναι απλό. Και στα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο. Από εκεί απορρέει το πρόβλημα. Στο χάρτη είπαμε, όταν εφαρμόζουν, γιατί θέλαμε να ακυρώσουμε μια ευρύτερη ερμηνεία του δικαστηρίου που έλεγε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα ίσχυαν στον τομέα του κοινοτικού δικαίου, in the field of the community law. Στις εξηγήσεις όμως του χάρτη προσπαθήσαμε να μαζέψουμε, να επανέλθουμε σε αυτό τον περιορισμό. Ε, όταν εφαρμόζουν ε, το κοινοτικό δίκαιο, τι σημαίνει αυτό. Όταν μεταφέρουν μια οδηγία ή όταν λαμβάνουν εκτελεστικά μέτρα για να εκτελέσουν ένα κανονισμό. Ακόμα και αυτό είναι σαφές ε, για τον πολίτη. Υπάρχει δράση της Ένωσης, υπάρχουν τα εκτελεστικά μέτρα των οδηγιών ή των εφαρμογής των κανονισμών. Τώρα, η δυσκολία που ανέφερε η συνάδελφος για τη Frontex απορρέει από την ερμήνεια που πάει ακόμα πιο μακριά σήμερα. Σε μια πρόσφατη υπόθεση που επιβεβαιώνει μια μακρά νομολογία, Σάιν Βίτλουνστάιν ονομάζεται, το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας εξηγεί τι σημαίνει εφαρμόζουν. Ήταν το θέμα ε, του αν η πριγκίπισσα του Λίχτενστάιν θα μπορούσε να καταχωρηθεί ως πριγκίπισσα ε, στην Αυστρία. Η Αυστρία λέει όχι, εγώ δεν αναγνώριζα τη Λουξεβγενία. Επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα με το καθεστώ της. Κανονικά είναι πρόβλημα της Αυστρίας. Ε, η Ένωση δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα για το τι καθεστώς έχει. Κάποιο στην Αυστρία. Η απάντηση του δικαστηρίου είναι όμω ότι αυτό φρενάρει την ελευθερία εγκατάσταση και κυκλοφορία τη πριγκίπισσα. Γιατί έχει ε, ένα τραπεζικό λογαριασμό που λέει πριγκίπισσα στη Γερμανία και ένα τραπεζικό λογαριασμό στην Αυστρία χωρί το τίτλο πριγκίπισσα. Αυτό όμω είναι εμπόδιο στην ελευθερία κυκλοφορία τη. Επομένω, η έννοια του πεδίου εφαρμογή είναι πάρα πολύ ευρύ. Είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε σε αυτήν την περίπτωση εάν το δίκαιο τη Ένωση ισχύει ή δεν ισχύει και προκειμένου, το δικαστήριο εφάρμοσε το χάρτη και την αρχή της ισότητας που υπήρχε στο χάρτη που έλεγε ο... η Αυστρία έχει δικαίωμα να ε, απορρίψει τον τίτλο. Είναι περίπλοκη η κατάσταση γιατί σε σχέση με τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι πολίτες δεν έχουν αφιβολίες. εφαρμόζεται πάντα σε όλες τις περιπτώσεις αλλά όχι ο χάρτης όμως. Είναι φυσιολογική αυτή η σύγχυση. Είμαστε σε ένα σύστημα πολλαπλών επιπέδων. Θα θυμάστε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αρχικά το, δι... το δίκαιο που εγγυόταν από το, από το ε, σύμβαση αφορούσε μόνο ε, απέρε μάλλον από την Ομοσπονδία. Πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Από πάνω. Δηλαδή, να κάνουμε όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά χρειάστηκε ο πόλεμος ανεξαρτησίας για να φτάσουν εκεί οι Αμερικάνοι. Και να πούμε, ο χάρτης ισχύει και στην Ένωση και στα κράτη-μέλη σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν χρειάζεται τέτοιος πόλεμος στην Ένωση. Αλλά θα έπρεπε να θεωρηθούν οι συνθήκες για να έχουμε αυτή την καθολική εφαρμογή του χάρτη. Μπορούμε λοιπόν να βγούμε από το... τη δυσκολία από κάτω προς το παρόν. Ε, από κάτω. Έχουμε πολλές πηγές. Εγώ θα έλεγα να συνεχίσουμε να καταχωρούμε με σαφήνεια για τον πολίτη ποιο είναι το περιεχόμενο των δικαιωμάτων και τι σημαίνει. Σε μία ιστοσελίδα σοβαρή, επαγγελματική και προσπελάσιμη να πούμε το δικαίωμα με ιδιοκτησία στο χάρτη σημαίνει αυτό συμπληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, προσθέτει αυτά και αυτά τα στοιχεία αυτή η σύμβαση και για, αυτά τα, για αυτό το δικαίωμα έχουμε λοιπόν ένα πανδέκτη πολύ συγκεκριμένο. Έτσι είναι πιο απλό. Τώρα, για το ε, πρόβλημα του πεδίου εφαρμογή. Στο βαθμό που είναι μία έννοια που θα υπόκειται πάντα σε νομολογιακή ερμηνεία, ποτέ δεν είναι απόλυτη σαφήνεια. Υπάρχει μία λύση που είναι αυτό που κάναμε στη Frontex. Δηλαδή, για να είμαστε σίγουροι, το Κοινοβούλιο ζήτησε τα θεμελιώδη δικαιώματα να ισχύουν στη Frontex. Κάθε φορά δηλαδή που νομοθετούμε ε, να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε με σαφήνεια ότι εφαρμόζεται η χάρτα, ο χάρτης ή δεν εφαρμόζεται. Δεύτερον, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα αφήνει κανένα παραθυράκι, κανένα κενό θα πρέπει ε, να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο όταν λαμβάνουμε ένα αίτημα από ένα πολίτη να εξετάζουμε την αίτηση αυτή και να λέμε δεν είμαστε εμείς αλλά είναι ας πούμε ο... στη Γαλλία ας πούμε εκείνος που υπερασπίζεται αυτά τα δικαιώματα εκεί τα στέλνουμε και θα πρέπει εκείνος να δεχτεί να κάνει αυτή την προσπάθεια. Επίσης, ο υπεύθυνο στην Ισπανία για τα δικαιώματα των πολιτών, ας πούμε, ε, αποστέλει τα αιτήματα στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όταν θεωρεί ότι αυτά εμπίπτουν εκεί. Μπορούμε να έχουμε μία άτυπη συμφωνία που θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν τουλάχιστον ότι υπάρχει μια απάντηση σε αυτά τα δικαιώματα και ότι το αίτημά του δεν πέφτει σε μια τεράστια τρύπα όπου η Κομισιόν ή το Κοινοβούλιο απαντούν «Α, συγγνώμη, δεν είναι δική μας υπόθεση, ε, βρείτε τα μόνοι σας με την εθνική νομοθεσία». Όχι, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Δεν, λέμε, δεν μπορούμε να λέμε «Δεν είμαι εγώ ε, υπεύθυνο. Πηγαίνετε να δείτε τον κύριο Χ, τον κύριο Ψ. Αυτό θα ασχοληθεί με το θέμα σας. Και τέλος, υπάρχει μια περίπτωση όπου εφαρμόζεται γενικά ο χάρτης σε όλους τους τομείς σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης και των κρατών μελών. Είναι η διαδικασία των κυρώσεων που προβλέπει από προβλέπεται από τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης του χάρτη, και νομίζω ότι τελευταίως έχουμε κάνει τα στραβά μάτια. Μην σκεφτείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο με πλειοψηφία του, τρί, του εν τρίτου των μελών τη σε περίπτωση παραβίαση. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε λοιπόν να ενεργοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία παρότι πρόκειται για εθνικό δίκαιο και εθνικές αρμοδιότητες. Αυτά και γράψει Πρεζιντέντε. Thank you very much to... Uh, εμείς σας ευχαριστούμε για αυτές τις τόσο αξιόλογες ε, εισηγήσεις και τώρα αρχίζει η συζήτηση. θέλω κάτι να σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σχετικό. Εγώ είμαι συντονίστρια των Πρασίνων στην Επιτροπή των Αναφορών και ήταν το θέμα της ελευθερίας του τύπου το οποίο ζητούσαμε μια μέρα σε σχέση με τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Τα κριτήρια Κοπενχάγης ισχύουν μόνο για υποψήφια χώρα. Δεν έχουν σχέση με την Ένωση. Αυτό θεωρήθηκε και αυτό ε, σοκάρισε την Επιτροπή Αναφορών. Τέσσερις ομιλητές έχω στον κατάλογο ο Βίκτορ Μποστινάρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά τους διακεκριμένους καθηγητές για τις παρεμβάσεις, διευκρινήσεις τους που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι σημαντικότερες από τη δήλωση της Αντιπροέδρου κυρίας Ρέντινγκ. Γιατί, διότι οι παρεμβάσεις σας επιβεβαιώνουν ότι σήμερα το κενό μεταξύ των πολιτικών μας αρχών, των νομοθετημάτων μας, είτε είναι συνθήκες, είτε είναι χάρτης ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, η διαφορά λοιπόν μεταξύ όλων αυτών και της πραγματικότητας σε κάποια κράτη-μέλη ε, ε καμιά φορά είναι ενισχυτικά μεγάλη. Τώρα λοιπόν που ζούμε μέσα στην κρίση, όπως είπε και ο καθηγητής ΕΡΤ, θα πρέπει αυτά να τα δούμε ακόμα περισσότερο. Τώρα, στα πρακτικά, ε, το μόνο όργανο το οποίο μπορεί να φροντίζει για την εφαρμογή των ε, νόμων είναι η Επιτροπή της Βενετίας μέσα σε δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είδε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις σοβαρής παραβίασης του χάρτη θεωρούμε αλλά η Κομισιόν ε, λέει κάτι διαφορετικό το ένα είναι η ελευθερία των μιμιέ στη Ρουμανία ένα άλλο η, ο, νέα νομοθεσία για τα μιμιέ στην Ουγγαρία και τέλος το Ουγγρικό Σύνταγμα και σε κάθε περίπτωση από αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έλεγε λυπούμεθα πολύ αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Ε, θα πρέπει ο χάρτης να ε, μεταφερθεί στην Εθνική Νομοθεσία, στην οριζόντια, στα κράτη-μέλη. Στην περίπτωση του Γκρικού Συντάγματος, η Επιτροπή της Βενετίας αναφέρει στις 25-26 Μαρτίου τρέχοντος, με τη γνωμοδότηση υπαριθμών 614, Λένε λοιπόν ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 στο του χάρτη οι διατάξεις αναφέρονται στα θεσμικά όργανα φορείς και οργανισμούς της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη επαρκώς τις αρχές της επικουρικότητας και μόνο όταν εφαρμόζεται η ενωσιακή νομοθεσία. Προσθέτουν όμως η Επιτροπή της Βενετίας λέει στην παράγραφο 25 ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στη χάρτη την ίδια νομική ισχύ όπως αυτή που έχουν οι συνθήκες 6 παράγραφος 1. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο χάρτης ε, περιλαμβάνοντας τις γενικές του διατάξεις στο κεφάλαιο 7 έχει άμεση ισχύ στα κράτη-μέλη και υπερέχει σε σχέση με αντικρουόμενη εθνική νομοθεσία. Επίσης ε, ε, απαγορεύει εθνικά τη λήψη εθνικών μέτρων που είναι ασυμβίβαστα με τις διατάξεις του χάρτη και ρωτώ τους διακεκριμένους καθηγητές να μας το εξηγήσουν αυτό, να μας εξηγήσουν πού εφαρμόζεται ο χάρτης και πού θα πρέπει να ερμηνεύεται ως πολιτική δήλωση, πράγμα που εφαρμοζεται το χαρτης και που θα έλεγα με την Επίτροπο Ρέντινγκ, γιατί έχουμε ενισχυτικά προβλήματα ε, και πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο χάρτης και να αντιδράσει η Κομισιόν. Θα τηρήσω τον κατάλογο μιλητών και εγώ ε, είμαι στη σειρά τώρα. Ε, αναφερθήκατε πολλές φορές στο Κοινοβούλιο για το... υπήρχε το πρόβλημα του πολεοδομικού νόμου. Ε, στο άρθρο 7 της συνθήκης το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιδρά πρώτο και ακούσαμε με έκπληξη στην προηγούμενη Επιτροπή ότι η Επίτροπος Ρέντινγκ ε, το είπε αυτό ατομική βόμβα στη συνθήκη. Δεν πρέπει να βάζουμε ατομικέ βόμβες στις συνθήκες, αλλά μόνο άρθρα που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται. Δεν έχουμε ατομικέ βόμβες εμείς. Ποια είναι η σχέση λοιπόν μεταξύ του άρθρου 2 στη συνθήκη και του άρθρου 7 σε σχέση με τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα γενικότερα, όχι σε σχέση με κάποιες χώρες επιμέρους που έχουν δικές τους ερμηνείες. Εκεί είναι ε, η αρχή της επικουρικότητας που παίζει ρόλο. Τι πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο εδώ. Επίσης, δεύτερον, στην Επιτροπή μας, μαζί με το διαμεσολαβητή, μιλάμε για διαφάνεια πρόσβαση στα έγγραφα και όλα τα σχετικά. Και υπάρχει σαφές μήνυμα που έχει πολλές φορές ε, φύγει από το Κοινοβούλιο και δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά παραμελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θα ορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο χάρτη, η διαφάνεια, η πρόσβαση στα έγγραφα, η καλή διοίκηση, που επίσης συμπεριλαμβάνεται, αναφέρονται όλα αυτά. Δηλαδή δεν εφαρμόζεται αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη κοινωτική νομο, ε, νομοθεσία. Αυτή η ερώτηση απευθύνεται στο, στους εναπομείνοντες καθηγητές μας, γιατί η αντιπρόεδρος έφυγε. Τέλος, ε, ε, η επόμενη ερώτηση από την Ταϊάννα Wallis. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους ομιλητές σαφώς αρχίζουμε να φτάνουμε στο βάθος του προβλήματος. Είναι δύσκολο για μας το κοινοβούλιο αυτό, γιατί πολλές φορές τα δικαιώματα αυτά υπερδημοσιοποιήθηκαν. Τώρα όμως θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους πούμε ε, κάτι αρνητικό, ότι ναι, θεωρήσατε ότι έχετε δικαιώματα αλλά δεν έχει. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο για μένα ως βουλευτή. Η ιδέα ότι έχουμε δύο παράλληλους διάβλους μεταξύ πολίτη και κράτους, κράτους μέλος και μεταξύ πολίτη και ένωσης και δεν υπάρχει διασταύρωση, αυτό ε, δημιουργεί προβλήματα όπως αναφέρθηκε. Υπάρχουν οικονομικά δικαιώματα με βάση τις τέσσερι ελευθερίες που είναι, θεσπίζονται ε, σε οδηγίες και υπάρχει σύνδεση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Άρα λοιπόν υπάρχει ε, διασύνδεση και οι πολίτες ε, δικαιούνται να αναμένουν αντίδραση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. ιδιαίτερα όταν όπως ακούσαμε υπάρχουν περιπτώσεις ε, κακομεταχείρισης κρατουμένων κλπ. Και όταν λαμβάνονται μέτρα από τρίτες χώρες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διασύνδεση και γι' αυτό θα πρέπει να μην ε, πούμε ότι δεν υπάρχουν τα δικαιώματα αυτά και ως ε, δικηγόρος και ως πολιτικός εκπήρας μπορώ να πω ότι εμείς θα πρέπει να ε, επεκτείνουμε την νομοθεσία, όχι να την συρρυκνώνουμε. Ευχαριστώ, Νταϊάννα. Τέσσερις ακόμη ομιλητές θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Ε, θα ε, δώστε σύντομες απαντήσεις, γιατί έχουμε λίγο χρονικό 20-25 λεπτά. Ποιος θέλει λοιπόν να κάνει να δώσει τις απαντήσεις. Ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Ε, σε ό,τι αφορά το ρόλο των ε, θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταρχήν θα πρέπει να εξετάζονται στην πολιτική διαδικασία. Από εκεί αρχίζουν. Μετά, αν παραπονούνται και καταγγέλουν οι πολίτες ότι κάποια θεμελιώδη ε, ανθρώπινα δικαιώματα δεν διαφυλάχθηκαν επαρκώς στις πολιτικές διαδικασίες για τον α ή β λόγο, θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να προσφύγουν στο δικαστήριο και να ζητήσουν από το δικαστήριο να παρέμβει. Περιπλέκεται το θέμα όταν πάει κανείς στο ημεδαπό δικαστήριο ή σε ένα δικαστήριο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περίπτωση παραβίασης του χάρτη. Πιστεύω όμως ότι οι διασυνδέσεις είναι αναπόφευκτες. Αποτελούν μέρος του συστήματος. Η εθνική και η ενωσιακή νομοθεσία δεν είναι, διαχωρισμένη δεν είναι διαχωρισμένη μεταξύ τους αεροστεγός. Κάποιοι τομείς είναι εθνικοί, άλλοι είναι ευρωπαϊκοί και άλλοι συνενώνονται. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο και αυτή είναι η φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, σχετικά με την ιδιοκτησία, η ιδιοκτησία, η προστασία της περιουσίας, όπως είπα, προστατεύεται από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Ήδη υπάρχουν αυτά και προϋπήρχαν του χάρτη. Αυτή θα ήταν λοιπόν η απάντηση δική μου. Ευχαριστώ πολύ. Δύο απαντήσεις. Καταρχάς δεν υπάρχει κενό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Το πρόβλημα είναι να μάθουμε ποιος είναι ο καλός δρόμος για να προστατεύσουμε αυτά τα δικαιώματα. Δηλαδή η εθνική δικαιοδοσία και το Στρασβούργο ή η οδός του χάρτη και ενδεχομένω του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Το δύσκολο δεν είναι να πούμε στου πολίτες ότι δεν έχετε δικαιώματα. Το θέμα είναι να κατευθύνουμε τον πολίτη. Έχουν δικαιώματα οι πολίτε. Το θέμα είναι να τον κατευθύνουμε στο σωστό δρόμο. Δεύτερον, μιλήσαμε για αξίες και για το άρθρο 5. 7, συγγνώμη. Πρόκειται για προστασία σε περίπτωση εξαιρετική. Αλλά δεν είναι αλήθεια ότι τα κριτήρια της Κοπενχάγης δεν ε, υπησέρχονται σε περίπτωση σοβαρής και συνεχούς ε, παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στη Λισαβόνα βάλαμε τα κριτήρια της Κοπενχάγης στο άρθρο 2 για τις αξίες. Και σε περίπτωση παραβίασης των αξιών, αν το κράτος δεν είναι μέλος, δεν μπορεί να γίνει μέλος. Και αν το κράτος όμως παραβιάζει την, ε, τις αξίες, οι διαδικασίες του άρθρου 7 ε, ισχύουν και δεν είναι ταπεινωτικές. Η πρώτη διαδικασία σε περίπτωση απειλής είναι να εξετάσουμε την κατάσταση. Δεν είναι μια καταδίκη για το κράτος. Προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα και να δούμε πώς μπορούμε να το επιλύσουμε. Στο παρελθόν, ενώ δεν υπήρχε τίποτα, ήμασταν πάρα πολύ αυστηροί, ας πούμε, με την ε, Αυστρία, Πιο πρόσφατα όμως, ε, παρότι υπάρχουν ένα κάρο μέσα στη διάθεσή μα κλείνουμε τα μάτια σε όλα τα προβλήματα. Ευχαριστώ, μου άρεσε αυτή η απάντηση. Τέλος. Η επόμενη. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Yeah, with the risk. Ε, ρισκάροντας να κάνω τις... Επειδή ρισκάρω να επαναλάβω τις ερωτήσεις θα είμαι σύντομη. Βλέπουμε ότι η Κομισιόν και ε, άλλα θεσμικά όργανα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θεωρούν τρόπον να ότι έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και μπορούν να τα χαμηλώσουν λίγο, να τις χαμηλώσουν ε, ιδιαίτερα σε σχέση με τρίτες χώρες πολλές φορές πιέζουμε τους άλλους να τηρούν τις ε, αξίες μας ε, και τα κριτήρια της Κοπενχάγης και εμείς δεν τα παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Έχω υπόψη μου εδώ τον νόμο των, ε, της Ουγγαρίας για τα ΜΜΕ ή την Ιταλία κλπ. Ακούσαμε την Επίτροπο να μας λέει ότι πρέπει οι πολίτες να ξέρουν όταν χτυπούν στη λάθος πόρτα καθηγήτρια Γκίλντ μας είπε ότι υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων που θέλουν να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε περισσότερα πράγματα για τη γνώμη σας επ' αυτού, γιατί έτσι θα εφαρμόσουμε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι είμαστε σε λάθος δρόμο και θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε περισσότερο αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα που μας είπατε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ Μάργαρετ. Ε, δεν άκουσα τις ε, ομιλίες και ζητώ συγγνώμη ε, στους ομιλητές που δεν άκουσα. Καθηγητά Ζακ, συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση σας ε, της κατάστασης και πραγματι η Επιτροπή Αναφορών Συχνά ακούγοντα την διαφορετική άποψη τη Επιτροπής τονίζουμε την Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να υπογραφεί από όλα τα κράτη-μέλη. Σωστά αναφέρατε το άρθρο 6, το σεβασμό της δημοκρατίας, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτο δικαίου και μετά έχουμε και τι κυρώσει, το άρθρο 7. Μια φορά απειλήθηκε η κατάσταση αυτή όταν ε, ο, στην Αυστρία όταν ο Χάιντερ έκανε ε, συνασπισμό ε, με τους χριστιανοδημοκράτες και ε, προειδοποιήθηκε η Αυστρία σε σχέση με τις δεσμεύσεις της με βάση τη συνθήκη. Εμείς ζητήσαμε πολλές φορές η αρχή αυτή να τύχει σεβασμού και στους οικοπεδοφάγους στην Ισπανία ε, που τους αρπάζουν τα, τις περιουσίες ε, χωρίς να υπάρχουν ένδικα μέσα για να προστατευτούν η έφεση ή οτιδήποτε. Ή όταν πάει κάποιος από τη μια χώρα μέλος στην άλλη και ο γάμος ε, με ενδεχομένω το ίδιο, με άτομο του ίδιου φιλού δεν αναγνωρίζεται. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια λοιπόν συρρυκνώνεται, αποδυναμώνεται έτσι. Έχουμε επίσης και κάτι άλλο εντελώς παράλογο τις διακρίσεις επί τη βάση της Ιθαγένειας όταν πρόκειται για τη συμμετοχή σε κάποιες εκλογές σε κράτη-μέλη. Ένας Ισπανός που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, δεν μπορεί να ψηφίσει σε όλες τις εκλογές, μόνο σε πολύ περιορισμένες εκλογές και αυτό ε, επαναλαμβάνεται σε όλη την Ένωση. Αν, έχουμε, αν είχαμε αν έχουμε ευρωπαϊκή ηθαγένεια πρέπει να την ορίσουμε και πρέπει να ορίσουμε τα δικαιώματα που τη συνοδεύουν, την πλαισιώνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα για τους πολίτες. Η Κομισιόν από τη μία πλευρά λέει ότι ο χάρτης εφαρμόζεται μόνο όταν αφορά τα θέματα που καλύπτονται από τις οδηγίες και του κανονισμού. Το Συμβούλιο τον αγνοεί και όταν πρόκειται για τα θεμελιώδη θέματα που ε, ανέφερα εγώ, αλλά συνεχίζει το Κοινοβούλιο να ασκεί πίεση. Ποια, πώς απαντάτε. Δύο ακόμη μέλη ζητούν το λόγο. Θα τους δώσω το λόγο τώρα. Και μετά από το γραφείο του διαμεσολαβητή ε, ζητεί κάποιος το λόγο. Και από το, την οργάνωση την Ελληνική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Λάντφορντ. Χαιρετίζω το σεμινάριο. Εγώ είμαι δραστήρια πιο πολύ στην Επιτροπή Λίμπε παρά στην Επιτροπή ΠΕΤΗ, την Επιτροπή Αναφορών, μάλλον στις πολιτικές ελευθερίες. Εντυπωσιάστηκα από την παρέμβαση της Elspeth ε, Guild Πώς είναι δυνατόν να λέει κανείς ότι το άρθρο 4 του χάρτη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση του, της νομοθεσίας για το δίκαιο αφού έχουμε ε, μεγάλο σώμα για νομοθετικό, νομοθεσίας για το άσυλο όσο, όχι τόσο όσο θα θέλαμε προσπαθούμε τώρα να ε, κάνουμε νέα δέσμη νομοθετική Στη, ο κανονισμός του Δουβλίνου είναι και ενωσιακή νομοθεσία όμως ε, αυτή η διασύνδεση ας πούμε, που ανέφερε η Νταϊάννα, οι τομείς ε, σύμπτωση και επικάλυψης, ε, αδιαμφισβήτητα ισχύουν εν προκειμένου. Πρέπει ο χάρτη να ισχύει στο, στην νομοθεσία για το άσυλο. Και βέβαια με πολύ ενδιαφέρον άκουσα την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα για τη Βρετανική υπόθεση ΕΝΕΣ. Υπάρχει και απόφαση από το Δικαστήριο του Στρασβούργου που λέει ότι δεν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, από το Βέλγιο αν θυμάμαι καλά ήταν κάποιοι. Ε, επίσης, ε, παράδοση και βασανιστήρια. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είχαμε αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καμία. Υπάρχει έκθεση που έχει παρουσιαστεί πάρα πολύ καλά και από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εγώ ήμουν αντιπρόεδρος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τέσσερα χρόνια. Ε, τίποτε. Ε, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί σιγή απόλυτη. Ενώ πρόκειται για πολύ σοβαρές παραδιάσεις και της ε, σύμβασης και του χάρτη εις ό,τι αφορά δηλαδή τη συνενοχή σε βασανιστήρια. είναι σαφή η περίπτωση. Πρέπει να μα απασχολήσει και να μα προβληματίσει όλου. Εις ό,τι αφορά τώρα το νόμο για τα ΜΜΕ, εθνικά συντάγματα κλπ. Και πάλι υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα να εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 7. Όμω η Κομισιόν λέει ότι ίσως υπάρχουν κάποιες τεχνικοί τομείς για την οδηγία για τα οπτικοακουστικά αλλά δεν αντιμετωπίζει το βασικό θέμα, την υπονόμευση των αξιών για να πω το λιγότερο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και σε τελευταία ανάλυση βλέπουμε αυτή την επιμονή αυτών των διπλωματών, αυτή τη διπλω, αυτής της διπλωματικής κουλτούρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και κράτη-μέλη και άλλοι φορείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρνούνται να καταπιαστούν με παραδιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας και των βασικών αξιών. Δηλαδή λες, δρούν λες και είναι κάποιο διακυβερνητικό φόρουμ. Δηλαδή πραγματικά είμαστε σε αμηχανία γιατί δεν θέλουμε να αλληλοκατηγορούμεθα. Ευχαριστώ. Και τέλος. Κύριο Σούκου. Ευχαριστώ. Είμαι Ρουμάνος από την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Λυπάμαι που η κυρία Μπένοβα δεν είναι εδώ, γιατί θα μπορούσε να μου απαντήσει. Αλλά τέλος πάντων, μπορώ να απευθύνω το ερώτημά μου προς υπόλοιπους. υπόλοιπου. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουμε μια νομοθεσία που ανανεώνει την ιδέα της ε, συλλογικής ενοχής. Ένα κράτος όπως η Σερβία που δεν είναι κράτος μέλος ψήφισε ένα νόμο θα έκανα ε, και ένα ερώτημα στην κυρία Μπένοβα για το γλωσσικό νόμο, αλλά και, την, και το Σόιεν, την, την υπόθεση Σόιεν. Ένας Ούγγρος που ήταν πρώην πρόεδρος της Ουγγαρίας, ε, τον σταμάτησαν στα σύνορα. Η ερμηνεία του θεμελιώδους στο χάρτη ήταν ενδιαφέρουσα. Η απάντηση ήταν ότι στην περίπτωσή του η ελευθερία κυκλοφορίας δεν ε, τέθηκε να αμφιβόλο διότι δεν είναι κλασικός πολίτης. Δεν είναι πολίτης όπως οι υπόλοιποι. Δεν είναι συνηθισμένο πολίτης. Έχουμε λίγα λεπτά για μία ακόμα ερώτηση. Σύντομη όμως, παρακαλώ. Είναι ο κύριος Ιαν Χάρντεν. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Ζήτησα το λόγο για να θέσω ένα ερώτημα στην κυρία Έλσπεθ Γκάιγκ. Μου έκανε εντύπωση η παρέμβασή της. Ανέφερε ότι ο Έλληνας διαμεσολαβητής είναι ενεργός για το θέμα των δράσεων των ελληνικών αρχών. Η Frontex είναι μια ευρωπαϊκή υπηρεσία και επομένως δεν ε, παίρνει εντολές από τον Έλληνα διαμεσολαβητή, αλλά ανήκει ε, στις αρμοδιότητες ε, του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Και επομένω τέτοια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Κυρία Γκάιντ, ξέρετε, λοιπόν, αν κάποια από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που ανησυχούν για αυτά τα θέματα σκέφτηκαν να στείλουν μία αναφορά στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τεζάουρο θα απαντήσει πρώτος από τους καθηγητές. Περνάμε τώρα σε απαντήσεις συνολικά. Θέλω να υπογραμμίσω ότι όταν μιλάμε για υπερβολικό ενθουσιασμό για το χάρτη της νίκαιας, είναι για να μην αποδυναμώσουμε το σύστημα ε, προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο χάρτης της νίκαιας ισχύει όταν ισχύει το κοινοτικό δίκαιο δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές. Οι περισσότερες περιπτώσεις ε, είναι αυτές. Επομένως, προσοχή. Βάζουμε κάποια όρια για να μην αποδυναμώσουμε το σύστημα. Δεν εννοούμε ότι δεν εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Αντίθετα, ε, στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζεται ο χάρτης. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν και μπορεί να ζητήσουν α, θεμελιώδη δικαιώματα σε τρία επίπεδα. Στο εσωτερικό, στο επίπεδο του Στρασβούργου και στο επίπεδο του Λουξεμβούργου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει Λουξεμβούργο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έπειτα υπάρχουν μια σειρά από δικαιώματα που δεν μπορούν να ασκηθούν παρά μόνο σε ενώπιον μη δικαστήριων. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Αλλά το πεδίο εφαρμογή του χάρτη της νίκης, δηλαδή του είναι αυτό του κοινοτικού δικαίου, γιατί ο χάρτης νίκης είναι κοινοτικό δίκαιο και αυτό... αυτός ο χώρος είναι τεράστιος. Δεν είναι περιορισμένος, είναι τεράστιος. Το πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυξάνει και θα αυξάνεται όλο και περισσότερο στο κοινοτικό σύστημα. Γιατί γιατί μόνο τα πρώτα χρόνια, για μια δεκαετία ας πούμε, το κέντρο βάρους του συστήματος ήταν τα οικονομικά θέματα. Δηλαδή ε, η κυκλοφορία των ε, εμπορευμάτων από όλες τις ε, τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες. Λίγο-λίγο όλα αυτά τα όργανα τα οποία προάγουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτό το κέντρο βάρους μετακινήθηκε προς την κυκλοφορία των προσώπων. Και πηγαίνει όλο και περισσότερο προς τα εκεί. Αυτή καθεαυτή την... Ε, δεν μιλάμε πια για τα οικονομικά θέματα και για την οικονομική διάσταση του ανθρώπου, για τον εργαζόμενο, για αυτό, ακόμα και για τον άνεργο, αλλά και για τους υπόλοιπους που δεν είναι οικονομικών, για τον φοιτητή, για οποιονδήποτε άλλον. Η κυκλοφορία των προσώπων μας έκανε να δούμε όλο και περισσότερο τα δικαιώματα του ανθρώπου και κυρίως τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όχι μόνο επεκτάθηκε ουσιαστικά επεκτάθηκαν τα δικαιώματα, αλλά κάλυψαν και μη κοινοτικούς πολίτες. Εγώ στο Ιταλικό ε, Συνταγματικό Δικαστήριο ασχολούμαι συχνά με θέματα μετανάστευσης και με μετανάστευση ανθρώπων εκτός κοινότητας. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και τους αναγνωρίζουμε τουλάχιστον τα θεμελιώδη δικαιώματα, Τουλάχιστον, αν όχι περισσότερο. Ίσως υπήρξε μια παρεξήγηση εδώ. Δηλαδή, ε, όταν εγώ είπα ότι ο χάρτης της νίκαιας πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή και να εφαρμοστεί με προσοχή. Σε καμία περίπτωση δεν είπα ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις. Όχι, εφαρμόζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Απλώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην αλλάξουμε τη φύση του και το πεδίο εφαρμογή του. Γιατί και γιατί η συνθήκη της ε, Λισαβόνας, τέλος πάντων η, συνθήκη της Νίκαιας και της Λισαβόνας έχουν κάποιες επιφυλάξεις, κάποια νεμένα αλλά για την εφαρμογή και την αύξηση των αρμοδιοτήτων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το κοινοτικό σύστημα βασίζεται σε μια ουσιαστική αρχή, κεντρική αρχή, που είναι οι, οι αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία και πολλές χώρες ενδιαφέρονται πάρα πολύ να εφαρμόσουν σωστά την αρχή των αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών. Παραδείγματο χάρη το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο κάθε τόσο τραβάει τα αυτιά για να φοβήσει τα παιδάκια. Sorry for being a little bit, but we are running out of time and I will give the floor now to... Πιέζει ο χρόνος, οπότε να δώσουμε αυτές αμέσως το καθηγητή. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδίω ευχαριστώ τον Ιαν για τα σχόλιά του αλλά και τις ερωτήσεις. Το πρώτο το οποίο θέλω να σας πω αφορά τον χάρτη. Ότι δηλαδή όπως ή οδήποτε μέτρο νομοθέτη με τα χρωματικά δικαιώματα είναι φορτισμένα πολιτικά αυτή η υπόθεση. Οπότε Δηλαδή βλέπετε ότι αυτή η προσδοκία να γίνεται δίκαιο, να γίνεται νόμος. Οπότε αυτό το έχουμε δει στο δικαστήριο επανειλημμένα. Οπότε υπάρχουν τα αντεπιχειρήματα ε, για, για τον σεβασμό της κοινωνικής ζωής κλπ. Σε σχέση με τα μέλη της οικογένειας, την αναγνώριση, τη θέσπιση κάποιων δικαιωμάτων. Δηλαδή να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν τα σχετικά δικαιώματα. Και βλέπουμε ότι Έχουμε δει κάποια παραδείγματα, κάποια προβλήματα για αυτά τα προβλήματα τα οποία εντείνονται όλα ένα περισσότερο γιατί η κατάσταση γίνεται όλα ένα και πιο δύσκολη κανείς δεν θέλει να προσβάλλει κάποιον και βλέπετε ότι το ΝΑΤΟ πολύ περισσότερο σε σχέση με την ε, Frontex δείχνει ευαίσθηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα οπότε τι να σας πω δεν ξέρω εάν ε, ε, ε, οι μη κυβερνικέ οργανώσει έχουν πλησιάσει τον δημοσιογραφητή. Πάντω, νομίζω ότι ε, αυτό ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ σωστό. Α, πάρα πολύ ευχάριστο το ότι το ΝΑΤΟ το κάνει αυτό. Δεν το περίμενα με τίποτα. Ελπίζω να έχετε δίκιο. Τέλο πάντων. Δεν ξέρω, πέστε μας αν έχετε τίποτε ιδιαίτερα σημαντικές παρατηρήσεις. Ναι, δύο την πρώτα Το αυτό πρώτο άρθρο 7 ναι, μα λέτε συνήθω δεν θέλει η Κομισιόν μα. Λέγω, μα κοιτάξτε κύριοι βουλευτέ, η συνθήκη τη αγώνα ε, προσδίδει σε εσά το δικαίωμα του να κινητοποιείτε την, ε, τη διαδικασία αυτού του άρθρου. Είδατε τι έγινε και με το Συμβούλιο. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό επομένως να μην επιτιθέμεθα, μην ρίχνουμε συνέχεια το, το, το, το φταίξιμο στην Κομισιόν να σκητάμε και το δικό μας περιβόλιο. Τι κάνουμε εμείς ήδη. βεβαίω και για το χαρτί ισχύουν αυτά. Φυσικά και το Βέλγιο, η, η Ελλάδα πρέπει να ε, τηρούν τα του άρθρου 4 και επίσης όσον αφορά τα ζευγάρια μου φιλοφίλων βεβαίως και αυτό έχει σχέση με την θερίδη ε, της ε, διακίνησης κυκλοφορίας με το χάρτη βεβαίως και έχουμε επίσης την οδηγία για το δικαίωμα διαμονής ε, όπου έχει κάποιες εσκίες όμως ε, νομίζω ότι ο χάρτης περιέχει αρκετά ευρείες διατυπώσεις ούτως ώστε να μπορούμε να εντάξουμε και να επιλύσουμε αυτά τα θέματα μέσω αυτού. Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όντως ε, θα, να δούμε, παρίσταται εδώ, εκπροσωπείται εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι νομίζω ότι την αφορούν διάφορα θέματα από αυτά που είπαμε τώρα. Σοφία Σπηλιοτοπούλου. Παρίσταται. Εκ του ελληνικού φορέα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί να λάβετε το λόγο, αν υπάρξει ο χρόνο, να απαντήσετε τι ερωτήσει, αλλά πάμε τώρα στο επόμενο πάνελ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ξεκαθρό όσο μας είπατε. Και περιμένω πώς και πώς να τα ξαναπούμε. Good Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Θα συνεχίσουμε τώρα τις εργασίες μα με το δεύτερο, όχι το τρίτο, το τρίτο πάνελ. Το θέμα είναι τώρα το πώ διακυπεριώνουμε τι καταγγελίε και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τι πρακτικέ που ισχύουν ει κάθε κράτο μέλο. Επομένω, τώρα θα ασχοληθούμε με τα φυσικά πρόσωπα, με την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους όποτε θεωρούν ότι έχουν εκείνα θυγή. Has been infringed and they think they should benefit from... Uh, όποτε έχουν φυγεί λέγω και θεωρούν ότι καλύπτονται από τον χάρτη. Shop The relief for individuals, rather than the... Αυτό είναι το θέμα του πάνελ, ξαναλέει ο Πρόεδρος. Όχι, δεν θα το δούμε από πολιτική πλευράς. Έχουμε βέβαια το άρθρο 7 το οποίο όμως βλέπει τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Θα ήθελα να σας πω ευθύ αμέσω ότι όποτε έχουμε να κάνουμε με δικαιώματα φυσικών προσώπων θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το δίκαιο των μαζών όποτε έχουμε ε, πάρα πολλέ υποθέσεις, αποφάσεις θα πρέπει να δούμε ποιος φορέας μπορεί αποτελεσματικά να επανορθώσει τα θυγέντα δικαιώματα οπότε θα πρέπει να δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει μέσω παντός διάβλου να εφαρμόσει τον ε, χάρτη ούτως ώστε να ωφελούνται όσο γίνεται περισσότερο τα φυσικά πρόσωπα. Ακούσαμε και από τους νομικούς στο προηγούμενο πάνελ. Ακούσαμε για τη λειτουργία των δικαστηρίων. Θα πρέπει να δούμε επίσης το πώς μπορούμε να έχουμε κάποιο αυτοέλεγχο των κρατικών δημοσίων φορέων. Οπότε θα πρέπει να δούμε επίση ότι εδώ πέρα υπάρχει ρόλο που μπορεί να διαρματίσει και ο διαμεσολαβητή, αλλά υπάρχουν και άλλοι εξωτερικοί τη Ένωση Φορεί. Για να δούμε τώρα, για να ταράξω τον έργο, πρώτα μια προκλητική ερώτηση. Δηλαδή, για πέστε μου, ποιο είναι το, το πιο αδύναμο, ο πιο αδύναμος κρίκος του συστήματος ούτως ώστε να αποκαθίσταται τα φυγέντα δικαιώματα και εγώ ω νομικό γνωρίζω ότι αν κάποιο το δικαιούται μπορεί ο δικαστή να αποκαταστήσει τα θηγέντα δηλαδή και τη ζημία που έχει υποστεί να μπορεί να πει ο δικαστή. ναι εγώ αποφασίζω κλπ κλπ κλπ οπότε και απονέμονται και πάλι τα θηγέντα δικαιώματα Όμω από την άλλη μεριά την άλλη μεριά τι αρμοδιό, τι προβλέπετε σε σχέση με τι καταγγελίε επίση, το δίκαιο των μαζών able to deal with effectively Ποιοι φορείς μπορούν να ασχοληθούν. Τι από πλάς ε, ποσοτική, από ε, βαθμό αποτελεσματικότητα, Τι γίνεται, τι γίνεται σε σχέση με τους κλασικού διάβλους που προβλέπονται και επίσης όσον αφορά την εφαρμογή του χάρτη, δηλαδή έχουμε την δικαιοσύνη, αλλά έχουμε και τα, τα, τα, τους φορείς αυτοελέγχου της διοίκησης των θεσμικών οργάνων. Πάμε για πέστε μας τώρα ποιοι ή μάλλον πριν προσφύγουν σε εσά οι παραπονούμενοι πού πάνε προηγουμένως έχουν πάει ήδη κάπου αλλού ή εσείς είστε ο πρώτος αποδέκτης των σχετικών παρμών των πολιτών και για πέστε μας σε σχέση με, τις, ε, με τους κλασικούς διάβλους, δηλαδή δικηγόρους, ε, δικαστήρια, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες δικηγόρων στην Ευρώπη. Τι γίνεται. Τι γίνεται επίση όσον αφορά τα πειθαρχικά και λοιπά συμβούλια που ελέγχουν την διοίκηση. Για πέστε μας επίσης σε πόσες περιπτώσεις νομίζετε ότι έχουν δίκιο οι παραπονωμένοι. Υπάρχουν κάποια όρια. Έτσι δεν είναι όσον αφορά το πόσο μπορεί να αποκαταστήσετε τα δικαιώματα. Επομένως, εδώ βρισκόμαστε εις μια διερευνητική αποστολή. Να διαπιστώσουμε το σύστημα, πώς λειτουργεί και πώς υλοποιεί τον χάρτη. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαγρυπνεί, ούτως ώστε να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό ο χάρτης υπέρ των ε, Ευρωπαίων. Και, όπως είπαμε και για άλλα πάνελ, κανένα όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί ατομικά να αποκαταστήσει κάτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί, δεν μπορεί ατομικά σε κάποιο συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο να αποκαταστήσει κάποια, κάποια ζημία. Πρέπει μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία παραβάση, η οποία όμω ποτέ από πλευρά νομικής άμεσα δεν απονέμει δικαιώματα ει φυσικό πρόσωπο. Και το ίδιο ισχύει, το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή των Αναφορών. Επιστολές, τέλο πάντων παρακλήσεις, εκκλήσεις, αλλά τελικά, τελικά τα πράγματα που καθιστούν τα δικαστήρια. Um, guests representing um, some of the specialized bodies for uh, Λοιπόν, οι προκεκλημένοι μας ε, εδώ εκπροσωπούν κάποια πάρα πολύ εξειδικευμένα όργανα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Πρώτα-πρώτα ο Ντομινίκ που είναι. έχει διατελέσει ευρωβουλευτής. Επί δύο θητείες. Και ο Ντομινίκ τώρα από τον Ιούνιο του 2011 είναι διαμεσολαβητής. Défenseur de droit in France. των δικαιωμάτων Défenseur de droit στα γαλλικά ή στην Γαλλία. Ντομινίκ Μανουέλ Αγγιλάρ Μπέλδα. Ισπανός. Είναι αναπληρωτής διαμεσολαβητής για θέματα παιδεία, κοινωνικής, πολιτικής και ασχολείται επίση με τις προσλήψεις από πλευράς του δημοσίου. Ντε Χόγκαν είναι αναπληρωτής διευθυντής της Επιτροπής του Φορέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ιρλανδία. Ο Πίτερ Ρέντιν επίσης είναι διευθυντής νομικής πολιτική, ισότητα και δεδομένων δικαιωμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σερβ Λεωνάρ ε, είναι νομικός σύμβουλος. Ε, ή στον ε, αρμόδιο για τα δικαιώματα των ελλήνων. Επίσης, ο δόκτωρ Ισραήλ Μπάτλερ που ε, ήταν πανεπιστημιακός προηγουμένως και τώρα ε, υπηρετεί στην κοινοτική υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχετε τώρα το λόγο και αν μπορείτε να αποπειραθείτε να απαντήσετε στα ερωτήματα τα οποία έθεσα στην αρχή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με καλέσατε σε αυτό το πάνελ, σε αυτή τη συζήτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσω στους ευρωβουλευτές και σε όσους συμμετέχουν σε αυτή τη συνεδρίαση ένα νέο όργανο, το οποίο δημιουργήθηκε στη Γαλλία μέσω μιας συνταγματικής μεταρρύθμισης. Δημιούργησε τον λεγόμενο υπερασπιστή των δικαιωμάτων, όπως τον αποκαλούμε, που είναι ένα όρος που θα υπάρχει τώρα και στο Σύνταγμα και συγκεντρώνει τέσσερα, ε, συγχωνεύει τέσσερι φορεί που υπήρχε πριν, το διαμεσολαβητή, τον όμπουτσμα δηλαδή της ε, Γαλλική Δημοκρατίας, τον υπερασπιστή των παιδιών, που ασχολείται με την καλή εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των παιδιών, την ύπατη αρχή καταπολέμησης των διακρίσεων και, την και υπέρ της προώθησης της ισότητας και τέλος την Επιτροπή Δεοντολογίας για την Ασφάλεια, που ασχολείται με τη δεοντολογία των επαγγελματιών της ασφάλειας, των σορφωνιστηρίων, της φυλακής, συγγνώμη, των της αστυνομίας, της χωροφυλακής κτλ. Ήταν τέσσερις ανεξάρτητοι φορείς που σήμερα ε, συγχωνεύονται σε έναν φορέα, σε αυτόν τον υπερασπιστή των δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά τη διοντολογία για την ασφάλεια, τις, τα δικαιώματα των παιδιών κτλ. Όλα αυτά, ε, για να μην τα ξεχνάμε, έχουμε ένα μηχανισμό που προβλέπει ότι ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων ε, έχει τρεις βοηθούς. Έναν που ασχολείται με τα παιδιά, ένα δεύτερο που ασχολείται με την καταπολέμηση των διακρίσεων και ένα τρίτο που ασχολείται με τη δεοντολογία των επαγγελμάτων τη ε, της ασφάλειας. Και διάλεξε τρεις γυναίκες που είναι βοηθοί μου. Υπάρχουν επίσης και τρία σώματα που ασχολούνται με τα παιδιά, τις διακρίσεις και την ε, διοντολογία των επαγγελματιών της ασφάλειας. Ο νομοθέτης έφτιαξε αυτή την ε, αρχιτεκτονική λίγο περίπλοκη, αλλά που λειτουργεί καλά τελικά, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε μία από τις αποστολές που παλιότερα εξασφαλιζόταν από μια ανεξάρτητη αρχή ή φορέα, να μην την ξεχνάμε. Ε, θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο μου ζητήσατε να σας δώσω κάποια νούμερα για να σας μιλήσω για δραστηριότητά μας. Πέρυσι, ε, πριν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης δηλαδή, τα τέσσερα αυτά όργανα είχαν, λάμβαναν περίπου 100.000 αναφορές ή παράπονα. Και ε, είχαν περίπου 80.000 πήγαιναν για την ε, διαμεσολάβηση, τον ombudsman, δηλαδή τον διαμεσολαβητή, περίπου 15.000 πήγαιναν, ε, ήταν υπόθεση αυτών που ασχολούνταν με τις διακρίσεις, περίπου 3.000 ε, για, αφορούσαν την ε, υπεράσπιση και την προστασία των παιδιών και 250 και 300 αφορούσαν τη διοντολογία στον τομέα της ασφάλειας. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι σε ένα τόσο τεράστιο τομέα οι 250 αναφορές ό,τι αφορά τη διοντολογία στον τομέα της ασφάλειας ξεχνόνταν από τους 80.000, λόγω των 80.000 φακέλου που λάμβανε ο διαμελασσολαβητής. Χάρη λοιπόν ε, στους βοηθούς μου και στο σώμα αυτό που δημιούργησα γύρω τους, ε, κάθε μία από τις αποστολές αυτές δεν λησμονείται. Λοιπόν, τώρα έχουμε τρεις άξονες ε, στην αποστολή μας. Καταρχάς, διεκπεραιώνουμε τους φακέλους. Εν συνεχεία, όλες τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας και τη διάδοση των καλών πρακτικών ειδικά στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, ε, μη απρόσκοπτη μάλλον πρόσβαση ε, στην απασχόληση, στις υπηρεσίες κτλ. Και η τρίτη δράση είναι οι προτάσεις μεταρρύθμισης που κάνουμε εμείς είτε προς την κυβέρνηση είτε προς το κοινοβούλιο. Αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα, μια ιδιαίτερη σημασία για το πολίτη γιατί το σύστημα πλουστεύεται. Προηγουμένως, όταν ένα άτομο, μια οικογένεια Φερρυπίν, είχε μια δυσκολία, γιατί δεν μπορούσε Φερρυπίν να γράψει το παιδί της που ήταν ανάπηρο, ας πούμε, και είναι σε καροτσάκι αναπηρικό, ε, δεν μπορούσε να το πάει εύκολα στο σχολείο. Ε, ασχολούνταν, θα μπορούσε να απευθυνθεί στον διαμεσολαβητή ή θα μπορούσε να απευθυνθεί στην αρχή που ασχολείται με την καταπολέμηση των διακρίσεων αντίον των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκε ή στο, σε αυτόν που ασχολείται με την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Γιατί μιλούμε για παιδί. Μερικέ φορέ ε, απευθυνόταν και στου τρει φορεί και λάμβανε διαφορετικέ απαντήσει και αντιφατικέ μερικέ φορέ. Τώρα έχουμε ε, ένα παραλήπτη και εμεί στο εσωτερικό μα διαλέγουμε την ε, καλύτερη διαδικασία, την πιο ενδεδειγμένη για να ικανοποιήσουμε όσου απευθύνονται προ εμά. Η μεταρρύθμιση είναι υπέρ του πολίτη γιατί η πρόσβαση πλέον είναι πιο εύκολη. Παλιότερα ο διαμεσολαβητή, θα έπρεπε κάποιο για να απευθυνθεί σε αυτόν να απευθυνθεί πρώτα μέσω ενό βουλευτή. Επίση για την διοντολογία για θέματα ασφάλεια το ίδιο ήταν. Έπρεπε να απευθυνθεί πρώτα κάποιο, ο ενδιαφερόμενο, σε ένα ευρωβουλευτή. Σήμερα οποιοδήποτε, ακόμη και ένα ε, ανήλικο, μπορεί κατευθείαν να απευθυνθεί στον στο σώμα αυτό που λέγεται η πράσπιση των δικαιωμάτων. Ειδικά στον τομέα της διοντολογίας ε, για την ασφάλεια, είχαμε, έχουμε περίπου 15 αναφορές στο μη. Είχαμε 15 αναφορές και τώρα έχουμε πάνω από 50. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπήρχε αυτό το φίλτρο των βουλευτών μερικές φορές δεν έστελνε ας πούμε, παραπάνω, στο παραπάνω επίπεδο α, τους φακέλους. Έκρινε ότι δεν είναι απαραίτητο. Σήμερα όμως κάθε περίπτωση, το κάθε πρόβλημα, κάθε αναφορά ε, έχει απρόσκοπτη, περνάει μέσα ένα απρόσκοπτο διάβολο και φτάνει ως εμάς. Ε, τα σώματα αυτά στους τρεις τομείς που ανέφερα έχουν σημαντικό ρόλο γιατί ε, εξηγούν τις αποφάσεις του υπερασπιστή για όλα τα νέα θέματα. Μου ζητήσατε προηγουμένως να σας πω αν υπάρχουν κάποιες διαδικασίες πριν φτάσει κανείς στον υπερασπιστή για την υπεράσπιση των παιδιών μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτε απευθεία σε εμά. Για την διοντολογία των επαγγελμάτων ασφάλεια το ίδιο. Για την καταπολέμηση των διακρίσεων επίση. Απλώ ζητάμε σε εκείνου που θέλουν να προσφύγουν σε εμά γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα με τη δημόσια διοίκηση να απευθυνθούν πρώτα ε, στη σχετική υπηρεσία ε, να κάνουν μια πρώτη προσφυγή εκεί. Και αν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, αν δεν λαμβάνουν καμία απάντηση, τότε ο πολίτης, όποια και αν είναι η εθνικότητά του, όλοι οι πολίτες, είτε διαμένει μόνιμα ή όχι στην ε, γαλλική επικράτεια, όλοι οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν σε εμά. Το ποσοστό επιτυχίας, μας ρωτήσατε ποιο είναι. Περίπου τα δύο, τα δύο τρίτα των φακέλων τελεσφορούν. Αλλά μιλάμε για τις παραδεκτές αναφορές. Αν ένα άτομο, ας πούμε, έχει ένα πρόβλημα ε, με, γιατί ο σκύλος του γείτονα καυγίζει το βράδυ, γιατί ε, δεν έχει, έχει το πρόβλημα ύπνου και μιλάει για το δικαίωμα στον ύπνο, ε, όχι βέβαια. Ε, για τις υποθέσεις που είμαστε αρμόδιοι, στις δύο τρίτες έχουμε, ε, στα δύο τρίτα των περιπτώσεων αυτών υπάρχει επιτυχία. πώ ε, φτάνουν σε εμά οι αναφορές, ε, είτε ταχυδρομείο κλασικό είτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ε, όπως καταλαβαίνετε, όλο και περισσότερο οι αναφορές ήταν ε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω email δηλαδή. Ε, φτιάχνουμε, ξαναφτιάχνουμε το εσωτερικό site του υπερασπιστή συχνά όταν οι άνθρωποι μας στέλνουν μια λεπτομερή επιστολή, μια ιδιόχειρη μάλλον επιστολή, συγγνώμη, ε, είναι πολύ πιο καλογραμμένες, πολύ πιο λεπτομερείς κτλ. Από ένα, από ένα email, ας πούμε, το οποίο είναι λίγο προχειρογραμμένο και εμβρασμό ψυχή συχνά. Ε, γι' αυτό του ζητάμε όλα τα στοιχεία. Ο δεύτερο τρόπο, στι πόλει, στι περιφέρειε, ε, στα διαμερίσματα, μπορεί να απευθυνθούν στου ε, προσώπους των τοπικών αρχών. Έχουμε 250 ε, επαγγελματίε στο Παρίσι και έχουμε 450 εκπροσώπους ε, σε όλη τη Γαλλική επικράτεια που είναι εθελοντές και που τους δίνουμε 350 ευρώ το μήνα ε, ένα μικρό ποσό. Ε, είναι νέοι συνταξιούχοι. Όλοι έχουν κάποια επαγγελματική εμπειρία. Κάποιοι ήταν αστυνομικοί, κάποιοι ήταν κοινωνικοί λειτουργοί, κάποιοι ήταν ε, του δικαστικού κλάδου, του, συγγνώμη, του νομικού κλάδου ε, και τους ενδιαφέρει αυτό που κάνουν. Κανένας δεν τους υποχρεώνει. Το κάνουν ε, δίνοντας, αφιερώνοντας τρεις μισές μέρες ε, σε, αυτό το, σε αυτή την προσπάθεια υποδεχόμενοι το κοινό. Αυτό ο μηχανισμός είναι πολύ σημαντικό. Συχνά όταν ο κόσμος έχει δυσκολίες με τη διοίκηση, ο πρώτος ε, λόγος του θυμού είναι ότι δεν συναντάνε ποτέ τον υπεύθυνο. Τους απευθύνουν ε, μέσω τηλεφώνου στον Άννα στον τον Καϊάφα, σε διάφορα ανώνυμα πρόσωπα, ενώ εδώ έχουμε 600 κέντρα υποδοχή σε όλη τη Γαλλία και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πίεση ήδη, γιατί ο κόσμο πάει κάπου τον, κάποιος τον δέχεται, τον σέβεται και τον ακούει. Ακόμα και αν στο τέλος δεν τους ικανοποιούμε, τουλάχιστον ε, τους αντιμετωπίσαμε ως πολίτες, με την πλήρη έννοια του όρου. Αυτός είναι ο πίνακα που ήθελα να σας παρουσιάσω για να απαντήσω στα ερωτήματά σας έτσι. Ευχαριστώ. Κύριος Μανουέλα Αγγιγέρ Βέδα. Ξεκινάω. Σας ευχαριστώ Ευχαριστώ εξ ονόματος του Ισπανού υπερασπιστή των δικαιωμάτων που μας καλέσατε να συμμετάσχουμε σε αυτό το σεμινάριο. Θα προσπαθήσω να περιγράψω τα χαρακτηριστικά της οργάνωσής μας. Το 1978 ξεκίνησε η διαδρομή αυτού του θεσμικού οργάνωση το οποίο υπηρετώ δυνάμει του, του άρθρου 54 ε, του σχετικού νόμου. Ε, ήταν ε, ένα νομοσχέδιο, νόμος τέλο πάντων του Κοινοβουλίου μας και υπερασπιζόμαστε όλα τα δικαιώματα ακριβώ αυτό που καλύπτει και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων. Σας έλεγα ότι δεν έχουμε τίποτα προηγούμενο. Είμαστε... Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο προηγουμένω. Ε, προερχόμασταν από δικτατορία και η πρόθεσή μα ήταν να προστατευτούν οι πολίτε ε, έναντι τη κακοδίκηση, α το πούμε. Και επομένω. Ε, το τότε η διοίκηση λειτουργούσε ως επικυρίαρχος και όχι στη βαστισότητα. Είμαστε ανεξάρτητο όργανο. Ε, τα τρία πέμπτα, δηλαδή μια ειδική πλειοψηφία κοινοβουλίου και γερουσίας μας ε, εκλέγει. Φασίζει για τον ορισμό μας τέλος πάντων. Ε, ε υπηρετούμε για μια θητεία ετή. και ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο έχει η υπηρεσία μας έχουμε ευρείες ερευνητικές αρμοδιότητες, μπορούμε να πάμε παντού, να ψάξουμε ε, στη, Οσνοφρατική διοίκηση, ε, ακόμα και στα, στα, στα μέρη, στα, στα έγγραφα τα απόρριτα και μπορούμε να διατυπώσουμε προτάσεις και συστάσεις προς την διοίκηση. Επίσης, έχουμε και εκτελεστική αρμοδιότητα. Ακριβώς όπως ε, έθεσε το ερώτημα ο Προεδρεύων για το κατά πόσον έχει αποδοτικότητα, έχει αποτελεσματικότητα η ρύθμιση ε, η οποία μας διέπει. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε δικαστικό όργανο. Άρα δηλαδή δεν έχουν ισχύ δικαστικών αποφάσεων οι συστάσεις μας. Όμως το 90% των όσων προτείνει ο διαμεσολαβητής υιοθετούνται, είναι αποδεκτές από την ε, διοίκηση. Δρούμε και σε επίπεδο αυτονόμων και διοικητικών κοινοτήτων της χώρας, σε τοπικό επίπεδο κλπ. Και, και όπως προείπα, το 80% των όσων προτείνουμε πιάνουν τόπο. Επίσης, κάθε χρόνο διεκπληρώνουμε 35.000 ε, καταγγελίες. 500 από αυτές προέρχονται από αυτεπάγγελτη έρευνα και άρα καταγγελία του ίδιου του διαμεσολαβήτου. Η ίδια πρωτοβουλία επομένω και μία έρευνα. Αλλά έχουμε και 18-20 χιλιάδες που προέρχονται από νομικά πρόσωπα, από ενώσεις προσώπων που θέλουν κάτι να καταγγείλουν συντάσσεται ετησίω μια έκθεση από την υπηρεσία μας. Εκεί εκθέτουμε τους προβληματισμού μα, τα θέματα που έχουν ανακύψει, ποιο συμμορφώθηκε, ποιο δεν συμμορφώθηκε, ποιος απάντησε, ποιο δεν απάντησε αυτά που είπαμε. Όλα όσα γίνανε εκθέτουμε εκεί. Και πέραν αυτών έχουμε και κάποιο είδους μονογραφικές εκθέσεις, δηλαδή που έχουν συγκεκριμένα έχουν συγκεκριμένο θέμα. Α πούμε όταν θέλουμε να, να, την προσοχή τη διοίκηση σε κάτι συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένο πρόβλημα, όπω α πούμε το φαινόμενο τη μετανάστευση που είναι κάτι καινούργιο για την Ισπανική κοινωνία, ξεκίνησε το 2000. Μιλάμε για εξωκοινωτικού που μέσα σε δύο χρόνια γέμισαν τη χώρα. Τι γίνεται επίση με την ε, παιδεία και αν καλύπτει τους ανήλικους μετανάστες, τη βία στα σχολεία, τι γίνεται με τα κέντρα όπου φιλοξενούνται οι πρόσφυγες και Επίσης ασχολούμεθα πάρα πολύ και με τη βία κατά ανηλίκων. Και επίσης με το, με το σοφρονισμό των ανηλίκων και τις σχετικές καταχρήσεις που γίνονται. Περιορισμό ελευθερίας ε, καταχρηστικό, ε, φαρμακευτική τους κάλυψη κλπ. Επίσης ε, μιλάμε για το ότι καλύπτουμε το τι γίνεται σε νοσοκομεία, φυλακές, σοφρονιστήρια ανηλίκων, αστυνομικά τμήματα και ονομάζεται υπηρεσία Εθνική Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, με διαπίστευση στον ΟΗΕ. Επίσης ασχολούμεθα και με την πρόληψη του βασανισμού. Αυτό δυνάμει νόμο του κράτους που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο. Επίσης μπορούμε να ελέγχουμε και την συνταγματικότητα κάποιων νόμων. Χρειάζεται να προσπογράψουν 50 βουλευτές, 50 μέλη της Γερουσίας που μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά ή επίσης μπορεί να το κάνει ο διαμεσολαβητής. Και αυτό επίσης είναι νόμος του κράτους από πλευρά ε, απόδοση σας είπα ότι το 80% των όσων λέμε πιάνουν τόπο. Ε, πολλές φορές έρχεται πρώτος σε εμάς ο πολίτης, δεν έχει πάει αλλού, δεν έχει διαμαρτυρηθεί στο, στην κρατική υπηρεσία. Λέει σε εμά κάντε εσείς αυτό το οποίο πρέπει. Καμιά φορά βέβαια συντρέχουν και κάποιες αποκλειστικές προθεσμίες. Άλλες φορές έρχονται κάποιοι αφού έχουν χάσει κάθε ελπίδα ενώ έχουν προσφύγει δηλαδή και αλλού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όσον αφορά το Δήμο της Μαδρίτης, τότε θέλαν να οικοδομήσουν ένα θέατρο, ε, άρχισαν τα έργα από την επιχείρηση και όταν ολοκληρώθηκε ε, το, το, η ανοικοδόμηση, η διπλανή πολυκατοικία ξαφνικά υπέστη τρομερές ρογμές τόσο πολύ που θα έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι. Γίνανε οι προσφυγές εκεί που έπρεπε, στο Δήμο κλπ. Είπαν ότι αυτό οφείλεται σε σεισμούς, ότι ήταν θέμα των υλικών, της των υλικών. Τέλος πάντων βρέθηκαν αυτοί άστεγοι κάποιοι που είχαν τα χρήματα προσέφηκαν στη δικαιοσύνη οπότε εμείς τότε είδαμε τι έγινε με την επιθεώρηση της αντοχής των υλικών τι έγινε τι, πώς ήταν πριν το κτίριο πριν βγουν αυτές οι ρογμές Οπότε και διαπιστώθηκε ότι αυτά οφειλόντουσαν στην ανοικοδόμηση αυτού του κτηρίου, αυτού του θεάτρου. Οπότε τότε ο Δήμος κατέβαλε σχετικές αποζημιώσεις και επεκατέστησε αυτούς που είχαν μείνει άστεγοι Οπότε ε, τελικά αποφασίστηκε να αποκατασταθούν οι ζημίες του κτηρίου που έμεινε ο κόσμος και κατόπιν να καταβάλει τα έξοδα η κατασκευαστική εταιρεία. Τώρα, κάτι το οποίο είπε εδώ ο συνάδελφος, τι γίνεται με το δίκαιο που διέπει τις, ε, τα ακίνητα στη, στην παραλία της χώρας μας. Στις ακτές εμείς οφείλουμε να εποπτεύουμε τη διοίκηση όσον αφορά την ομιμότητα των διοικητικών πράξεων. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να τροποποιήσουμε το κείμενο δίκαιο. Οπότε, εμείς προτείνουμε στα κόμματα και τους προτείνουμε ούτως ώστε εκείνοι να νομοθετήσουν και να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Οπότε υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, οπότε και καταλήγουμε στο να υπάρχει μια κατάφορη αδικία που νεφίσταται ο κόσμος. Οπότε και τώρα κάποια στιγμή θα φροντίσουμε το ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα αυτό. Είμαι στη διάθεσή σας αν έχετε τυχόν ε, ερωτήσεις, αν μπορώ να τις απαντήσω. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Προχωρούμε τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα ετοιμάσει μια παρουσίαση με PowerPoint, αλλά πρέπει να εξοικονομήσουμε χρόνο. Θα προσπαθήσω να κρατήσω το ενδιαφέρον σας, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση καταρχήν. Θα μιλήσω για θεσμικούς, θεσμικά όργανα σε εθνικό επίπεδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ακούσουμε και ομιλία για αυτό το απόγευμα. Αυτά, αυτοί οι οργανισμοί, οι ιδρύματα, είναι ανεξάρτητες οργανώσεις, χρηματοδοτούνται από το κράτος, έχουν θεσμική νομική ε, ε, ε, βάση, ε, λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Αυτό είναι σημαντικό. Η ανεξαρτησία θα πρέπει να διασφαλίζεται με καταστατικό κανονισμό ή το Σύνταγμα. Πρέπει να υπάρχει πλουραλισμός στα μέλη, να υπάρχει ευρεία εντολή που θα στηρίζεται στα ε, ε, καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς ε, παρέμβασης σε τοπικό, εθνικό, ε, περιφερειακό επίπεδο. Ε, η εντολή τους περιλαμβάνει νομοθετική εξέταση, σχέδια νόμου που υποβάλλονται σε επιτροπές κλπ. Έρευνα, κάνουμε δική μας έρευνα, εξετάζουμε πολιτικές, ποια είναι η πολιτική, ας πούμε και η διοικητική πρακτική την πρόθεση, προωθούμε ανθρώπινα δικαιώματα, εκπαίδευση, κατάρτιση. Πολλοί από εμά συμμετέχουν ε, στην εκπαίδευση όλων, από παιδιά σχολικής ηλικίας μέχρι ε, δημοσίους λειτουργούς. μου λένε, διακόπτει ο πρόεδρος, ε, να μιλάτε αργότερα, πιο αργά, ναι. Ε, για την προσφυγή τώρα έχουν διαφορετικές εντολές ε, τα, οι θεσμικοί αυτοί οργανισμοί αλλά δεν μπορούν να ε, παρεμβαίνουν στα δικαστήρια. Μπορούμε να κάνουμε έρευνες όμως, μπορούμε να χειριζόμεθα καταγγελίες. Έτσι λοιπόν τρόπον την κινούμεθα και ε, στο επίπεδο εθνικών και διεθνών προτύπων έχουμε και λειτουργίες που ξεπερνούν την απλή προσφυγή ε, και κοιτάζουμε και θέματα μεταρρύθμισης νομοθετικής κλπ. Υπάρχουν τέσσερις περιοχές όπου λειτουργούν τα ιδρύματα αυτά και ε, λειτουργούμε στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης όπου υπάρχουν 36 τέτοια ιδρύματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εθνικοί οργανισμοί, 22 έχουν καθεστώς βαθμίδα Α με βάση τις αρχές του, των Παρισίων. Οι 36 αυτοί αποτελούν το, ε, την Ευρωπαϊκή Ομάδα των Εθνικών Ιδρυμάτων 15 ε, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 18 τέτοια ιδρύματα, 12 έχουν καθεστώς Α και θα σας πω ποια είναι. Είναι η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βόρεια Ιρλανδία, ε, Σκοτία, τρεις επιτροπές. Υπάρχουν πέντε που έχουν καθεστώς Β, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, ένα η Ρουμανία με καθεστώς Σ και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 11 κράτη-μέλη της Ένωσης που είτε έχουν ένα θεσμικό όργανο που διαπιστεύεται ή δεν διαπιστεύεται ή δεν έχουν τέτοιο ίδρυμα. Χαρακτηριστική εντολή ε, του καθεστώτος Α ασχολείται με ε, πολιτικά ε, δικαιώματα, δικαιώματα του πολίτη, οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε κενά στην εντολή. Εξετάζομαι λοιπόν και το Σύνταγμα και τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών. Η Αντιπρόεδρος ε, Ρέντινγκ σήμερα το πρωί μίλησε για την ε, σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών ε, Διεθνών Θεσμικών Οργάνων πολλές φορές χρησιμοποιούμε αποφάσεις των δικαστηρίων εμείς στα εθνικά αυτά ιδρύματα. Για να μπορούμε να ε, συμπράττουμε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πρέπει να είναι σημαντική υπόθεση γιατί είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι, οι ικανότητές μας περιορισμένες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, τι σημασία έχει ο χάρτης για το συγκεκριμένο έργο μας και ήδη ο προηγούμενος ομιλητής από την Ισπανία μίλησε για αυτά τα θέματα κακή μεταχείριση των ε, ε, μεταναστών, ε, οικονομική πρόσφυγη, καταστάσεις, συνθήκες στις φυλακές, κακοποίηση παιδιών, ανθρώπων με αναπηρία. Αυτά τα βλέπουμε κάθε μέρα και τα αντιμετωπίζουμε με τον δικό μας τρόπο ε, και ο χάρτης βέβαια θα πρέπει να εφαρμόζεται, αλλά θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη καθοδήγηση για το τι μπορεί να γίνει. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους βουλευτές εδώ, ε, θα έλεγα ότι εμείς παρουσιαζόμαστε μπροστά σε επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών για να δώσουμε στοιχεία για το πώς χειρίζονται τις υποθέσεις στις χώρε μας ως εθνικά όργανα. Ε, πολλές φορές ε, πρέπει να πάμε σε επιτροπές, κάναμε κάποιες εργασίες για την παράδοση ατόμων και εμφανιστήκαμε, εμφανιστήκαμε και στην προσωρινή επιτροπή που είχε συστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Τώρα, τα εθνικά ιδρύματα μπορεί να είναι εθνικές επιτροπές, μπορεί να είναι φορείς ισότητας, μπορεί να είναι ο ε, και λειτουργούν με βάση τις συμβάσεις για τη βασανιστήρια κλπ. Δεν είναι όλοι οι διαμεσολαβητές ε, τέτοια ιδρύματα. Ο Ισπανός βέβαια ε, διαμεσολαβητής μπορεί να συμβάλλει στην μεταρρύθμιση της νομοθεσίας. Γι' αυτό είναι και καθεστώτος Α. Ο Πολωνός, ο Ισπανός, διαμεσολαβητής, η Ιρλανδική Επιτροπή μπορούν να έχουν ε, διευρυμένες δραστηριότητες. Θα ήθελα να πω επίσης ότι κάναμε μία έρευνα πριν από την παρουσίαση αυτή ως ομάδα για να ε, σας δείξουμε τι καταγγελίες παίρνουμε και πώς τις χειριζόμεθα. Όπως είπα πριν μπορούμε επίσης να έχουμε νομική ε, προσώπηση ανθρώπων, Ιρλανδική Επιτροπή. Μπορούμε να είμαστε αμήκους κούριε στη Σκοτική Επιτροπή είναι παράδειγμα. Μπορούμε να παρουσιαστούμε στην ε, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το κάναμε αυτό κάποια στιγμή σε μια υπόθεση στήρωση ε, κοριτσιών. Καμιά φορά τα ιδρύματα έχουν διπλή εντολή, μπορούν να πάνε μόνο σε υποθέσει ισότητα ε, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο και στη Δανία που είναι καθεστώτο Α. Κάποια εθνικά ιδρύματα, γιατί καλύπτουμε πάρα πολλού τομεί, πολλέ φορέ θα πρέπει να έχουμε διακριτική ευχέρεια για να δούμε δηλαδή, για να αποφασίσουμε ποιε καταγγελίε θα χειριστούμε και χρειάζονται κατευθυντηρίε γραμμέ για όλα αυτά. Κάποια ιδρύματα έχουν περισσότερες ε, λειτουργίες εντολής στα πλαίσια της μεταρρύθμισης νομοθεσία, όπως στη Γαλλία. Τα εθνικά ιδρύματα που δεν χειρίζονται τέτοιε καταγγελίες, παραπέμπουν αλλού, όπως στη Δανία έτσι γίνεται. Μπορούμε να παραπέμψουμε δηλαδή ανθρώπους σε εφορείς ισότητας, νομικής βοήθειας, στο διαμεσολαβητή, σε υπεύθυνου ε, για την προστασία δεδομένων. Είπε και ο πρόεδρο ότι αναγνωρίζουμε ότι τα δικαστήρια μπορούν να ε, δώσουν λύση. Ε, μια δυσκολία είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν εξοδικαστική λύση, δεν θέλουν δηλαδή να δαπανίσουν τόσα χρήματα στα δικαστήρια και να φτάσουν και μέχρι το Στρασβούργο. Κάποια εθνικά ιδρύματα μπορούν να το κάνουν αυτό, Πολωνία, Ισπανία. Συχνά προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που αρχίζει να κάνει τώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να δει δηλαδή κάποιες τάσεις, ε, να δει συστημικά ζητήματα και να τα χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε να δούμε την υποκείμενη διοικητική πρακτική στις φυλακές ή σε ε, ε, φιλόφιλους κλπ. Ε, συμπεραίνοντας λοιπόν κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι αυτά τα εθνικά ιδρύματα που εξετάζουν καταγγελίες πολλές φορές δεν έχουν δυνατότητα να παρέμβουν πολύ στα πλαίσια της εντολής τους όσοι δεν ε, χειρίζονται καταγγελίες ε, περισσότερο ασχολούνται με θέματα μεταρρύθμισης νομοθεσίας. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η αφύπνιση είναι θέματα που απασχολούν τους εθνικούς τα θεσμικά όργανα αυτά, τα ιδρύματα, αλλά πολλές φορές ε, δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα αυτά. Είναι μια συνεχιζόμενη πρόκληση και για μας και για όλους σε νομικές υποθέσεις μπορούμε να παρεμβαίνουμε και παρουσιαζόμεθα μπροστά στα εθνικά ή διεθνή δικαστήρια. Τέλος, είμαστε ανοιχτοί ε, σε διάλογο, σε συζήτηση. Πιστεύουμε ότι είναι ε, μια αμφίδρομη διαδικασία. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έρθει να μας πει ότι πρέπει να εφαρμόζουμε το χάρτη. Πρέπει να υπάρχει ευαισθησία και σε σχέση με τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικά ιδρύματα και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Thank you very much uh, for... Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Serge Leonard. Πάμε στον ε, Serge Leonard. Serge Leonard, Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Είμαι εκπρόσωπος της ε, Νομικός Σύμβουλος της Γαλλικής Κοινότητας ε, του Βετγίου. Να σας παρουσιάσω λίγο το, το φορέα μου που δημιουργήθηκε το 1991 μαζί με την επικύρωση τη Διεθνή για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Είναι ένας ε, φορέας που είναι τμήμα της κυβέρνησης της γαλλικής κοινότητας, της γαλλόφωνης κοινότητας, συγγνώμη, αλλά έχουμε την υποχρέωση ανεξαρτησία σε σχέση με, το, με την κυβέρνηση. Ποια είναι η αποστολή μα. Καταρχά, έχουμε μια αποστολή ενημέρωση ό,τι αφορά τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Έχουμε μια ε, δουλειά δηλαδή πρόθεση αυτή τη σύμβαση. Έχουμε μια αποστολή ε, εξακρίβωση τη σωστή επαλήθευση του νόμου. Έχουμε μια αποστολή ε, συστάσεων προ τι διάφορε κυβερνήσει στο Βέλγιο ε, οργανώνουμε ομάδες εργασίες για συγκεκριμένα θέματα. Μπορεί να αφορούν ε, την επικύρωση της σύμβασης της Χάγης του 1996 που αφορά μια σειρά από θέματα. Έχουμε επίσης μια αποστολή να συλλέγουμε ε, ατομικές αναφορές, ατομικές καταγγελίες. Σε σχέση με το τελευταίο αυτό, σε σχέση με αυτό το σημείο θα μιλήσω σήμερα, γιατί γι' αυτό μας καλέσατε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη μας ε, είναι ότι είμαστε ένας φορέας της ε, γαλλικής ε, κοινότητας. Η, το Βέλγιο είναι μια πολύ περιπλοκή χώρα και τα, το θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών είναι οριζόντιο θέμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση σε σχέση με τη διαχείριση των ε, καταγγελιών που διεκπεραιώνουμε. Ε, πρόκειται για καταγγελίες που προέρχονται από ιδιώτες και που αφορούν το πεδίο ε, αρμοδιοτήτων της γαλλικής κοινότητας ε, ε, έχουμε κάποια προνόμια σε σχέση με αυτές. Έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε την πρόσβαση σε φακέλους και να ζητήσουμε να μας τυπώσουν τους φακέλους, να καθορίσουμε προθεσμίες και να πάμε σε όλα τα κτίρια τα οποία επιχορηγούνται από τη γαλλική κοινότητα. Έχουμε κάποια προνόμια λοιπόν. Αυτά τα προνόμια τα χρησιμοποιούμε όμως πολύ σπάνια. Στα κείμενα έχουμε τα προνόμια, ε, αυτά τα όπλα, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε στην πραγματικότητα. Υπάρχουν μια σειρά από τομείς και θέματα που αφορούν το Ομοσπονδιακό κράτος, γιατί το Βέλγιο είναι περίπλοκη χώρα, σας το είπα. Υπάρχουν οι κοινότητες, υπάρχουν οι περιφέρειες και υπάρχει και το Ομοσπονδιακό κράτος. Και όλα αυτά τα θέματα τα διαχειρίζεται το, και το Ομοσπονδιακό κράτος. Ε, τα δικαιώματα του παιδιού, ας πούμε, υπάρχει και εκεί αρμοδιότητα. Πρέπει να ξέρετε ότι στο Βέλγιο τα μέτρα προστασίας που αφορούν τους ανήλικους εγκληματίες ή τους ανήλικους που έχουν βρίσκονται σε κίνδυνο, τα παίρνει το δικαστήριο. Αλλά την εφαρμογή αυτών των μέτρων, ε, τοποθέτησης, ε, συνοδείας των παιδιών κτλ. Ε, είναι αρμοδιότητας της γαλλικής κοινότητας. Υπάρχουν λοιπόν κάποια οριζόντια θέματα και πρέπει να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε αυτά τα θέματα. Να δώσω ένα παράδειγμα, ένα άλλο παράδειγμα. Την ε, διεθνή οθεσία. Έχουμε δύο κεντρικέ αρχέ. Έχουμε μια κεντρική αρχή ομοσπονδιακή που είναι επιφορτισμένη να επαληθεύει την ε, ισχύ των εγγράφων, αν υπάρχει συνένεση ε, και αν ενισχύει, αυτή, είναι, ε, αυτή η συνένεση και έχουμε και μια κεντρική αρχή που ασχολείται με την ε, έγκριση, με την ε, ε, συνοδεία. Ε, μερικές φορές με τις απαγωγές των, των γονέων, ας πούμε, ασχολούμαστε και με αυτά. Ε, έχει να κάνει με την προστασία των παιδιών. Γι' αυτό η γαλλική κοινότητα ασχολείται με το θέμα αυτό που έχει μια διάσταση που αφορά την προστασία ο φορέας μας συνεργάζεται με άλλες αρχές, με άλλους φορείς που δεν ανήκουν στη γαλλική κοινότητα, δεν είναι αρμοδιότητα της γαλλικής κοινότητας. Θα ήταν αδύνατο να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα, χωρίς όμως να προσφύγουμε σε άλλους φορείς, ε, να ζητήσουμε τη βοήθεια άλλων φορέων. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια ολόκληρη προσπάθεια εδώ, ε, να οργανώνουμε συνεδριάσεις, ε, να διατηρούμε επαφές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Δεν είναι πάντα εύκολο φυσικά, γιατί όταν έχετε φορείς του ομοσπονδιακού κράτους, το θεσμικό πρόβλημα το ξέρετε. Ξέρετε ότι οι φορείς έχουν μια τάση να λειτουργούν σαν επαγγελματική συντεχνία. Ο καθένας θέλει να διατηρήσει τα προνομιά του. Αυτό είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα μια νεαρής κοπέλα, η οποία αποτέλεσε, που την εγκατέλειψαν εδώ στο Βέλγιο, ο ο πατέρας της είχε άδεια διαμονή στην Αγγλία, την εγκατέλειψαν εδώ στις Βρυξέλλες, ε, ο πατέρας φεύγει με τα έγγραφα, επιστρέφει στην Αγγλία, δεν υπάρχουν πια έγγραφα. Για αυτό το θέμα λοιπόν εξετάσαμε τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 56 του κανονισμού του, Βρυξελών, του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Οργανώσαμε μία συνεδρίαση με, τους, ε, με τις κεντρικές αρχές, με με τους εισαγγελείς και με τις αρχές που είναι υπεύθυνε για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Αλλά τίποτα δεν μας δίνει αυτό το προνόμιο. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία. Πρόκειται για την ηθική αρχή που έχει ένας φορέας. Αν και ο όρος είναι λίγο υπερφύαλος. Πήραμε λοιπόν, εν πάση την πρωτοβουλία για να δράσουμε έτσι. Φυσικά, έχουμε και άλλες αποστολές ένας φορές ο δικός μας ε, δίνει συμβουλές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο κόσμος χρειάζεται ενημέρωση. Ένα από τα καθήκοντά μας είναι να ενημερώνουμε. Ε, ερχόμαστε σε επαφή για να ενημερώσουμε και να δώσουμε και συμβουλές. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε άτομα που γνωρίζουν ε, τα τις διεθνούς προστασίας των παιδιών, τις διεθνούς προστασίας των νέων, άτομα λοιπόν καταπτυσμένα χρειαζόμαστε. Επίσης, στα πλαίσια της αποστολή μας, έχουμε μια παράπλευρη αποστολή, που απορρεί από την αποστολή της παροχής συμβουλών, ε, είναι το καθήκον του προσανατολισμού. Έρχονται διάφορα άτομα που να μας δουν, ε, παιδιά ή έφηβοι. Συχνά όμως ε, τα αιτήματα, οι καταγγελίες απορρέουν από τους γονείς τους ή από τους συγγενείς τους ή τους γνωστούς τους. Πρέπει να τους ε, κατευθύνουμε, να τους πούμε προς τα πού να πάνε. Αυτό είναι σημαντικό. Για το ερώτημα που μας θέσατε, Πρόεδρε, τώρα. Ο φορέας μας είναι ο, ένας φορέας τελευταίας προσφυγής, ας πούμε, τελευταίας καταφυγής. Κάποιο ε, φτάνει σε εμά όταν έχει εξαντλήσει μια σειρά από δυνατότητε. Ε, δικαστικέ προσφυγέ, διοικητικέ προσφυγέ. Φυσικά συχνά τα άτομα δεν γνωρίζουν τα όργανα της ε, γαλλικής κοινότητα, Ε, εάν δεν τα ξέρουν, τους προσανατολίζουμε προς αυτά, προ τα κατάλληλα όργανα, προ του κατάλληλους φορείς. Είμαστε δηλαδή μια υπηρεσία στην οποία καταφεύγει ο πολιτή ε, στο τέλο. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των δράσεών μας, Έχουμε μια, συνοδή, μια επιτροπή έτσι, πλαισίωσης, αλλά δεν έχουμε αποτιμήσει ποσοτικά τα νούμερα. Η προστασία, η προσπάθεια, ο αγώνας προστασίας του παιδιού είναι ένας καθημερινός, μόνιμος, αέναος αγώνας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ και πολλά χρόνια πολεμάμε κατά της εγκατάλειψης του σχολείου, και της αποτυχίας στο σχολείο στα, στη γαλλική κοινότητα. Έχουμε πάρα πολύ κακά ποσοστά ή πολύ κακού βαθμούς ας πούμε. Εδώ και δέκα χρόνια πολεμάμε αυτό το, αυτή τη μάστιγα. Η κυβέρνηση πήρε θέση και είπε θα προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε ε, την, την τάση που υπάρχει στη γαλλική κοινότητα να αφήνουμε τα παιδιά στην ίδια τάξη έγιναν ε, μελέτες από τον ΩΣΑ και τα λοιπά και από άλλους ε, φορείς για το θέμα αυτό, για το πρόβλημα αυτό. Δεν μπορώ να σας πω ότι ήμασταν πολύ αποτελεσματική. Χρειάστηκε 10 χρόνια να πολεμήσουμε. Έπειτα θα ήταν πολύ επιρμένο εκ μέρους μας να το πούμε αυτό. Δεν είμαστε εμείς οι νικητές ε, αυτού του αγώνα. Υπάρχει μια σειρά από οργανώσεις γονέων που προσπάθησαν, που κινήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Το θέμα λοιπόν της αξιολόγησης. Έχουμε μια επιτροπή πλαισίωσης και μας εποπτεύει τρόπον την αυτή επιτροπή. Ευχαριστώ, Πίτερ Ρέντινγκ, τελευταίος. Καλημέρα. Ακόμα μέρα είναι, πρωί είναι, καλημέρα. Θα σας παρουσίαζα μια ωραία παρουσίαση με PowerPoint, αλλά φαίνεται ότι η τεχνολογία μας ε, εγκατέλειψε και έτσι θα τα παρουσιάσω με τον καλύτερο τρόπο. Ήθελα να σας μιλήσω για πέντε κεντρικά ζητήματα σχετικά με το πώς χειριζόμεθα καταγγελίες για ανθρώπινα δικαιώματα. Καταρχήν, ποιες είναι οι βασικές μας λειτουργίες και καθήκοντα, πώς χειριζόμεθα τις καταγγελίες ε, εσωτερικά και αυτό τι συνέχεια δίνεται και πώς ε, επιλύουμε στρατηγικά τις διαφορές, γιατί υπάρχει ένας τρόπος παροχής υποστήριξης και βοήθειας στα άτομα. Τέταρτον, θα σας πω ε, ποια είναι τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουμε και ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε στη δουλειά μας στο μέλλον, γιατί πολλά από τα θέματα αυτά έχουν αντίκτυπο και σε άλλους φορείς ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Τέλος, τι συμπεράσματα μπορούμε να αντλήσουμε ίσως από αυτά τα θέματα. Καταρχήν η Επιτροπή μας είναι καταστατικός ανεξάρτητος φορέας όπως και άλλα θεσμικά εθνικά ιδρύματα που φροντίζουν για θέματα καλών σχέσεων και ισότητας και λοιπά στην κοινωνία. Είμα, έχουμε καθεστώ καθιστός α όπως είπε και ο Ντέσμοντ και είμαστε ε, λειτουργούμε από τον Οκτώβριο του 2007. Ίσως ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε μία σειρά ε, αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων ε, στα οποία πρέπει να ανταποκρινόμεθα, να δίνουμε συμβουλές και υποστήριξη στα άτομα με διάφορους τρόπους, θα έρθω και σε αυτό μπορούμε να ε, χειριστούμε θέματα επίλυσης διαφορών παρεμβαίνοντας σε κύριες υποθέσεις, μια φορά ως αμίκους κιούρεϊ, ε, μπορεί καμιά φορά να κινήσουμε διαδικασία με το δικό μας όνομα, εμείς αυτοδικαίως δηλαδή, όταν υπάρχει, θεωρούμε θέμα παραβίασης χωρίς να υπάρχει προσφεύγων, μπορούμε επίσης να κάνουμε έρευνες σε επιμέρους τομείς και αυτό είναι σημαντικό για μας, διότι ε, όπου εντοπίζουμε συστημικά προβλήματα, οι έρευνες είναι σημαντικός τρόπος ε, για να διασφαλιστούν κοινωνικές αλλαγές. Ε, κάναμε έρευνες πρόσφατα και κάνουμε έρευνες σε θέματα παρενόχλησης σε ανθρώπους με αναπηρία αυτό συνιστά έγκλημα κατά των αναπήρων. Κάνουμε επίσης έρευνα σε σχέση με την αντιμετώπιση ανθρώπων ηλικιωμένων και αναπήρων που είναι στο σπίτι και ε, σε θέματα εμπορίας ανθρώπων στη Σκωτία. Ένα βασικό πρόβλημα, και αυτό έχει να κάνει με τα εμπόδια, είναι ότι δεν έχουμε την εξουσία να εκπροσωπήσουμε άτομα σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σε περιπτώσεις διακρίσεων όπου εκεί μπορούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα εμπόδιο και θέλουμε να παρακάμψουμε το εμπόδιο χρησιμοποιώντας άλλες εξουσίες με τρόπο δημιουργικό εξουσίες που διαθέτουμε. Σε ό,τι αφορά το πώς χειριζόμεθα τις καταγγελίες, υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι όπου τα άτομα και οι οργανώσεις μπορούν να έρθουν και να προσφύγουν σε μας. Έχουμε ένα helpline, γραμμή βοήθειας, ε, που είναι σημείο εισόδου για όλες τις ε, ερωτήσεις και καταγγελίες και έχουμε 50 ανθρώπους προσωπικό που βοηθούν εκεί. Αυτό συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε σχέση τώρα με τις οργανώσεις ή ε, νομικές εταιρείε κλπ, τους ενθαρρύνουμε να έρχονται σε επαφή με τη νομική μας ομάδα, γιατί μπορεί και εκείνοι να μας αναθέσουν να δουλέψουμε πάνω σε ένα θέμα ή να δουλέψουμε πάνω σε μια υπόθεση. Έχουμε επίσης λεπτομερείς συμβουλές στο ε, στην ιστοσελίδα μας ε, ε, αναφορές στο χάρτη πως μπορούν να γίνουν οι προσφυγές και οι καταγγελίες και που μπορούν να προσφύγουν οι άνθρωποι αν δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Ένα παράδειγμα ας πούμε, που δεν, σας είπα ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε άτομα, μπορούμε να τους πούμε ποιες άλλες οργανώσεις μπορούν να βοηθήσουν, μπορεί να είναι οι διαμεσολαβητές, μπορεί να είναι ε, κάποιες ομάδες ε, νομικών. Ένας άλλος σημαντικός τομέας που έχει να κάνει με την παροχή βοήθειας είναι ότι έχουμε ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων ε, ύψους 10 εκατομμυρίων στερλινών που δώσαμε σε 100 οργανώσεις περίπου που παρέχουν νομική βοήθεια και άλλες συμβουλές, καθοδήγηση, ανατολισμό σε θέματα ε, ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν δεν μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς, μπορούν άλλοι. Τους παραπέμπουμε σε αυτούς. Κάποια νούμερα τώρα, στατιστικά, δεν τα βλέπετε, θα σας τα πω εγώ. Ε, σε ό,τι αφορά τον αριθμό καταγγελιών που παίρνουμε, από το Helpline, τη γραμμή βοήθεια, τα τελευταία 3,5 χρόνια ε, είχαμε 5.600 ε, καταγγελίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι κάποιες ομάδες φαίνεται να καταγγέλουν πιο συχνά. Δεν κάναμε ανάλυση για να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά για παράδειγμα 469 ήταν οι καταγγελίες από ανάπηρα, ε, ανάπηρους και 364 από εθνικές μειονότητες, ενώ μόνο 16 καταγγελίες είναι από ομοφιλόφιλους και 6 δια, φιλο, φιλομεταβατική. Θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση για να δούμε γιατί δεν έρχονται και δεν κάνουν καταγγελίες σε εμάς αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, εις ό,τι αφορά ε, τα θέματα που, των καταγγελιών, ως επιτοπλίστων πρόκειται για κεντρική δια, κυβέρνηση, τοπικές ε, κυβερνήσεις, ΟΤΑ, αστυνομία, ε, δικαστήρια, ε, ειρηνοδικεία, το σύστημα υγείας και έχει νόημα. Δηλαδή εξηγείται αυτό γιατί ε, είναι κάποιοι βασικοί τομείς αυτοί που εκεί μπορούν να υπάρξουν προβλήματα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρίτον, τρίτος τομέας. Πώς χειριζόμεθα την επίλυση διαφορών στρατηγικά. Ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι είναι πολλές οι καταγγελίες και δεν μπορεί κανείς να τις χειριστεί όλες, άρα πρέπει να είναι επιλεκτικός. Ε, θα εστιάσουμε στα σημαντικά και τα σημαντικά ε, πρέπει να αποφασιστούν από τα δικαστήρια. Έχουμε λοιπόν μια στρατηγική επίλυση διαφορών που θέτει το τομεί προτεραιότητας. Για φέτος ε, είναι η καταπολέμηση τροπομοκρατία, η αστυνόμευση, οι διαμαρτυρίε, πολύ σημαντικό θέματα ιδιωτικής ζωής, εμπορία. Ε, περικοπή δημοσίων δαπανών ε, που πλήττουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν είναι μόνο μεγάλο θέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των υποθέσεων όπου συμμετείχαμε, ε, σε 63 παρεμβάσεις στη χώρα, 16 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δύο παρεμβάσεις κάναμε στα ευρωπαϊκά εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δύο ε, παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η μία ήταν ε, η υπόθεση Κόλμαν για άτομο με ειδικέ ανάγκες, με αναπηρία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα αναφέρω όμως μια πρόσφατη υπόθεση που αφορούσε το χάρτη και που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί δείχνει Πώ οι φορείς ισότητα και ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να, έχουν, να παίξουν ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ερμηνεύοντας το χάρτη. Ε, αυτή είναι η υπόθεση ΕΝΕΣ ε, εναντίον του Υπουργού Εσωτερικών. Η, η αναφορά είναι ΣΥΓ κάθετος 411 τέσσερα κάθετος 10 είναι η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα από 22 Σεπτεμβρίου φέτος. Είναι πρόσφατη υπόθεση και είναι πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση διότι αφορά το δικαίωμα ασύλου και τους κανονισμούς που θεσπίστηκαν το 2003, ο 343 του 2003, που είναι ο νόμος που προβλέπει ότι η αίτηση ασύλου θα πρέπει να κρίνεται στη χώρα της πρώτης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε εκείνη τη χώρα που ήρθε, μπήκε. Οι κοινικοί θα πούνε ότι αυτό έγινε για να μην πάνε σε χώρες ε, οι αιτούντες άσυλο όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι κοινικό αυτό. Είναι γεγονός. Έτσι συμβαίνει όντως. Η υπόθεση είναι σημαντική γιατί εξέταζε το θέμα ενός Αφγανού ετούντος άσυλο που ήρθε στην Ελλάδα και μετά προχώρησε μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο και ζήτησε άσυλο εκεί, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκείνος έλεγε ότι η αίτησή του θα έπρεπε να κρυθεί όχι στην Ελλάδα αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί αν επέστρεφε στην Ελλάδα οι συνθήκες ε, για τους ετούντες άσυλο είναι τόσο κακές που υπάρχει η περίπτωση να παραβιαστεί το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, το δικαίωμα ε, στην αίτηση ασύλου κλπ. κλπ. Τώρα, ο Γενικός Εισαγγελέας εξέτασε... Α, ένα άλλο θέμα που ετέθη ενώπιον του δικαστηρίου ήταν το πεδίο εφαρμογής του πρωτοκόλου 30, που είναι το πρωτόκολλο το οποίο η Βρετανική και Πολωνική κυβέρνηση ε, συμφώνησαν μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία του χάρτη. Και το θέμα ήταν ο χάρτης έχει πλήρη ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς αυτό έχει τεράστια σημασία για οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά το χάρτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχει και επιπτώσεις και για τους φίλους στην Πολωνία. Δεν λειτουργεί το PowerPoint, δεν μας βοηθάει η τεχνολογία ακόμα. Ε, έγιναν λοιπόν παρεμβάσεις δικές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και ο τη Αρμοστία για τους πρόσφυγες και η Διεθνή Αμνηστία παρενέβησαν, οπότε αυτό σας δίνει να καταλάβετε τη σημασία ε, αυτών των υποθέσεων. Επίσης είναι σημαντικό ότι το δικαστήριο αναφέρθηκε σε μια πρόσφατη απόφαση, την MSS, κατά του Βελγίου και της Ελλάδας, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εξέτασαν παρόμοια υπόθεση, αλλά ε, ήταν κάποιο που έφτασε στο Βέλγιο, αλλά αρχικά πέρασε από την Ελλάδα και αν θα είχε δυνατότητα να ζητήσει άσυλο στο Βέλγιο. Εκεί έκριναν ότι παραβιάστηκαν ανθρώπινα δικαιώματα βάσει του άρθρου 3 αν επέστρεφε δηλαδή θα υπήρχε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του βάσει του άρθρου 3. Για να, να μην μακρηγορώ, η έκβαση, ή τουλάχιστον η γνωμοδότηση, γιατί περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου, είναι το, ε, ε, δικαστήριο είπε ότι δεδομένων των ανησυχιών ε, στην Ελλάδα ε, θα πρέπει να εξετάσει το Ηνωμένο Βασίλειο εάν παραβιάζονται δικαιώματα κατά την επιστροφή. Δεν ήταν λοιπόν αυτόματη υπόθεση, δηλαδή δεν εστάλει αυτομάτως πίσω. Αυτό λοιπόν σημαίνει και αν η απόφαση είναι προς αυτή την κατεύθυνση ότι η Βρετανική κυβέρνηση και άλλα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάζουν αν οι αιτήσει θα πρέπει να κρυθούν στη δική του τη χώρα και όχι στην Ελλάδα, εάν η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, δεν τελείωσα. Πολύ σύντομα ε, για τα εμπόδια. Πολύ σύντομα. Είπα ότι δεν μπορούμε να δώσουμε ε, υποστήριξη σε άτομα. Για πολλά εθνικά ιδρύματα ένα πρόβλημα είναι οι περικοπές στη χρηματοδότηση. Θα γίνουν περικοπές κατά 50% τον επόμενο χρόνο στους προϋπολογισμούς μας. Επίσης υπάρχουν απειλές ε, σε σχέση με την αντίληψη που υπάρχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τέλος θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και ένα θέμα ε, για το αν ε, οι φορείς ισότητας στα εθνικά ιδρύματα μπορούν να παρεμβαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν συμμετείχαν στην, ε, κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης από το Εθνικό Δικαστήριο. τώρα η απόφαση είναι ότι δεν μπορούν. Και αυτό αντιφάσκει στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπου οργανώσεις σύμφωνα με την οποία μη κυβερνητικέ οργανώσει και οργανώσει σαν τη δική μα μπορούν να παρεμβαίνουν. Οπότε εδώ έχουμε ένα πρόβλημα στο σύστημα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στη λειτουργία του. Και μάλιστα μίλησα και με το γραμματέα του Δικαστηρίου και συζητώ και με ε, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει περισσότερο την Ένωση δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας του χάρτη και του ρόλου των Εθνικών Ιδρυμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σταματώ εδώ και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα είπατε και ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριο Μπάτλερ όσον αφορά αυτό το πάνελ τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόσφατα έμαθα ότι κάποιο ξεκίνησε ένα κόμμα που το λέει το κόμμα κατά του PowerPoint. Να δούμε τι θα, θα βγάλουν οι βουλευτέ. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τρία ειναι πρώτα πρώτα με μια γενική έποψη του θέματος των καταγγελιών στα κράτη-μέλη. Κατόπιν θα μιλήσουμε για πληροφόρηση από τα δικαιώματα και κατόπιν να δούμε πώς καλύτερα θα καλυφθούν τα θύματα από αρμόδιους φορείς. Δύο τινά θα ήθελα να σας πω. Πρώτα-πρώτα για τις δεσμενείς διακρίσεις. Έχουμε να κάνουμε με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις σχετικές καταγγελίες και δεύτερον έχουμε κάποια στατιστικά και θα έπρεπε να έχουμε από, από πολλά στοιχεία, από πολλά, πολλούς που ασχολούνται με την εισόδο και τις δεσμένες διακρίσεις. Τα στοιχεία εδώ μας δείχνουν ότι έχουμε τρομερή ποικιλία και διαφορά μεταξύ των κρατών μελών στο πόσες υποθέσεις καταγράφονται. Πολλές χιλιάδες σε κάποια κρατημέλη, σε άλλα εκατοντάδες, σε άλλα λιγότερες από 20 ή 10 υποθέσεις. Αυτό είναι το 2010. Αλλά τα ίδια είναι και το 2009. Εμείς κάναμε κάποιες ε, προσαρμογές όσον αφορά ε, τα στοιχεία σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας για να μπορούμε να ξέρουμε να έχουμε κάποια τάξη μεγέθους τι γίνεται επομένω ε, με τα μεγάλα κράτη, τι γίνεται με τα μικρά. Ακόμα όμως και με τέτοιου είδου προσαρμογή παραμένουν οι μεγάλες διαφορές σε σχέση με το πώ υποθέσει βγαίνουν πού. Άρα δεν εξηγείται αυτή η διαφορά μόνο από τον πληθυσμό της χώρας. Θα μπορούσε κανείς να δει τα πράγματα επιφανειακά και να πει ότι τα πάνε πάρα πολύ καλά τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν λίγες υποθέσεις. Εκεί, επομένως, έχει λίγες δυσμένες διακρίσεις κλπ. Μια άλλη μεριά, Γαλλία, Σουηδία κλπ. Ε, ε, δεν τα πάνε πολύ καλά γιατί έχει εκεί πολλές υποθέσεις. Αυτό όμως είναι αφελής, ερμηνεία και επιφανειακή. Το σωστό είναι να, να πούμε ότι εξηγείται το φαινόμενο αυτό από το πόσο ξέρει ο κόσμος τα δικαιώματά του. Το 2009 δημοσιεύθηκε μια έρευνα. Κατόπιν κάποιου γκάλωπ λέγαμε ότι ρωτήθηκαν 23.000 από μετανάστες ή από εθνότητες, του τέλο ξένης καταγωγής. Και τον τέταρτον εξ αυτών δεν μπορούσαν να, να δώσουν ούτε το ένα, ούτε ένα, ένα, όνομα, ούτε για έναν οργανισμό φορέα που ασχολείται με τις δημιουργίες διακρίσεις, την ισότητα κλπ. και όταν του ε, ονομάσαμε κάποιο τέτοιο φορέα το 60% αυτών είπαν δεν το έχουν ακούσει ποτέ το, το φορέα, το σώμα αυτό. Μόνο τον τέταρτον ήξεραν ότι υπάρχει, προβλέπεται προστασία για δεσμενείς διακρίσεις. Για απασχόληση, στέγαση κλπ. Άρα, δεν είναι μόνο θέμα του ότι δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν γιατί δεν ξέρουν ε, αν υπάρχει κάποιος τον οποίο μπορούν να προσφύγουν. Αυτό το πρόβλημα επίσης εξηγεί γιατί ε, πάρα πολλές περιπτώσεις που θα έπρεπε δεν καταγγέλλονται. Ο 2% είπε ότι ακόμα και αν έχουμε δεσμείς διακρίσεις προσεύγει μόλις το 20%. Άρα θα πρέπει να έχουμε όλοι περισσότερες υποθέσεις. Επομένως δεν, δεν έχουμε ακόμα επίγνωση της ε, τάξης πάντων, της τάξης μεγέθους. Τώρα, παράγοντες που αυξάνουν τη δυσκολία του να απευθύνει κανείς εκεί που πρέπει. Πρώτα πρώτα, σε πολλά κρατημέλη έχουμε πάρα πολλούς φορείς. είναι θέμα αρμοδιοτήτων. Ε, οι ανηλίκους ασχολούνται για άλλοι με βασανισμού κλπ κακοδιοίκηση. Επίσης, έχουμε διαχωρισμό ανάλογα με το αν κάποιες φορές ασχολείται περιφερειακά, τοπικά κλπ. Άρα κάποιος ο οποίος δεν ε, ξέρει, δεν ξέρει πού να απευθυνθεί. Πολλές φορές έχουμε και επικαλύψεις. Μεγαλύτερη σύγκριση φέρνει αυτό. Και πολλές φορές, ακόμη και να έχουμε πολλούς φορείς, υπάρχουν κάποια κενά στις, στην κάλυψη. Άρα κανείς μπορεί να πηγαίνει από εδώ από εκεί και να μην βρίσκει τη σωστή πόρτα να χτυπήσει. Τώρα, μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι τι γίνεται αν κανείς πηγαίνει και χτυπάει τη λάθος πόρτα. Αυτή τη στιγμή ε, κάνουμε μια μελέτη για αυτό το θέμα και βασιζόμαστε σε συντέξει από πολλά κρατημέλη, 200 θύματα δεσμενών διακρίσεων, και ενδιάμεσες οργανώσεις. Κάτι επί το οποίο απαντούν οι ερωτώμενοι είναι Μάλλον αυτό το ρωτούμε τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Αν έρθει κάποιο σε εσά και ήσασταν αρμόδιοι, θα το στείλετε αλλού. Υπάρχει επομένω τέτοιου είδους ανταπόκριση. Υπάρχουν οι εξή λύσει. Έτσι μπορεί τα θύματα να βοηθηθούν και να μπορούν να χτυπήσουν τη σωστή πόρτα. Μία δυνατότητα, το είπαν και οι άλλοι προελίσσαντε, είναι το να δούμε τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμα φτιάξουμε ένα, ε, ένα φορέα, ένα σώμα τέτοιο, ούτω ώστε να μην υπάρχουν κενά. Πόροι, αμεροληψία, αρμοδιότητες ερευνητικέ και δυνατότητα να επηρεάζεται η νομοθεσία και η πληροφόρηση. Όλα αυτά τα κριτήρια θα χρησιμοποιούνται για να χαρακτηριστεί ένας φορέας κατά πόσο είναι δόκιμος. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε λένε, και περισσότερου φορείς που ασχολούνται με τα φαινόμενα που συζητούμε έχουμε 12 φορείς τέτοιους σε 10 κράτη-μέλη. Τρεις φορείς είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο PowerPoint είχα έναν χάρτη που δείχνει πάρα πολύ όμορφα τι, ποιο είναι τι, αλλά δεν γίνεται να το δείτε. Και να δούμε τώρα ποια είναι τα πλέον εκτίματα. Αυτά τα ακούσαμε και τα στοιχεία λέει ο Πρόεδρος. Αν μπορείτε προχωρήστε στα συμπεράσματα. Καλά δεν σας πω τα στοιχεία. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι αν κανείς έχει ένα τέτοιο οργανισμό ε, εθνικού επέδου ξέρει κανείς που να πάει και επηρεάζεται επομένω και, και η νομοθεσία και έτσι τελικά έχουμε λιγότερες καταχρήσει. Βέβαια, όσο πιο λίγους φορεί έχουμε, τότε πιο πολύ τίνει το κράτος να κόβει τους φόρους. Οπότε, ίσω να έχουμε κάποιο είδου οργανώσει υποτύπων ομπρέλας και έτσι να υπάρχει μία πύλη, ας το πούμε, πάει κάποιος και από εκεί συντονίζεται το έργο όλων των επιμέρους φορέων. Αυτό είναι το υπέρ. Το κατά είναι ότι αν υπάρχει μία οργάνωση, αυτό δεν αποκλείτων υπάρχουν ακόμη κενά στο πλέγμα προστασίας. Μια οργανωση αυτο δεν τον υπαρχουν ακομη κενα δυνατότητα να υπάρχει προσέγγιση αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων. Όποιος και να πάρει την καταγγελία την διεκπεριώνει ή στέλνει εκεί που πρέπει το θύμα ε, δηλαδή έρχεται πάει κάποιος πάει μια πόρτα και το τον ακούνε και μετά τον ειδοποιεί αρμόδια αρχή δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα οι φορείς τα κάνουν όλα τέλος να υπάρχει ένα, ένα σημείο μόνο εισόδου στο σύστημα αυτό αυτό μπορεί να γίνει και με λογισμικό, μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε κάποιες ερωτήσεις με ένα πρόσωπο. Και έτσι τελικά ξεκαθαρίζονται τα πράγματα, είναι και διαδραστικά. Υπάρχει ένα σχετικό πρόγραμμα το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2013 και άλλη μια επιλογή είναι στο τέλος αυτής της διαδικασίας που είναι σχεδόν σε όλα τα στοιχεία Κατόπιν υπάρχει όλη η καταγγελία και διαβιβάζεται εκεί που πρέπει. Είναι μεγάλο τεχνολογικό άλμα αυτό. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει το σύστημα, όμως είναι εύκολο για το χρήστη. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορούν όλοι, δεν έχουν όλες τις τεχνολογικές γνώσεις για να κάνουν αυτό που χρειάζεται. Οπότε πάλι ξαναγυρίζουμε στην παραδοσιακή λύση της μη κυβερνητικής much. This was interesting. Now... Πάρα πολύ όλα αυτά και τώρα έχουμε τις ερωτήσεις. Τις ερωτήσεις από το κοινό. Mrs. Auken. Thank you very much, Mr. Chair. And... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους συζητητές για όλα τα ενδιαφέροντα που μας είπαν. Έχω τώρα κάτι να ρωτήσω. Τον Ισπανό διαμεσολαβητή. Ξέρετε ότι είσαστε ο καλύτερο πελάτη τη Επιτροπή Αναφορών. Τόσε και τόσε αναφορέ λαμβάνουμε από την Ισπανία. Μήπως θέει το σύστημα δικαίου που έχετε. Να σας αναφέρω τα θέματα που μας απασχολούν. Έχουν το θέμα αυτό με, τη, με τα εμπράγματα δικαιώματα στην, ε, στις παραλίες, στην ακτή της χώρας. Είναι πολύ ευθέρετο. Μπορεί δηλαδή κανένας ε, να πάει σε ένα δοχείο μου εκτισμένο πάνω στον γελό αλλά δεν μπορεί να έχει σπίτι του, το πήραν. Και νομίζω ότι είναι οικονομική η λόγη. Θυμάμαι στη Βαλένθια ιδίω ότι εκεί το ίδιο το δίκαιο που το οποίο ισχύει παραβιάζει ορμένα δικαιώματα. Μπάστε και το σύνταγμα. Και αν προσφύγουν σε δικαστήρια είναι πολύ έξοδες οι δίκες και κρατάνε τόσο πολύ. Άρα δεν έχουν βοήθεια. Τελικά ο περιφερειακός διαμεσολαβητής μας βοήθησε πολύ. πολύ. Ο διαμεσολαβητής της Βαλένθια. Άρα σας ερωτώ. Θεωρείτε ότι προστατεύετε τον κόσμο, προστατεύετε τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτως ώστε να μην, μπορεί κάποιος, να, να μην χρειάζεται κάποιος να προσφύγει στις κοινωνικές αρχές. Έχουμε άλλα λεπτά, λέει ο Πρόεδρος. Και έχω κι άλλη, κι άλλη ερώτηση, λέει κύριε Άουγκερ. Ναι, ναι, ναι, αλλά ίσως, ε, ίσως να μπορείτε να τα πείτε έξω, στο πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει κύριε κυρία Okay, so... One short comment and two... Ένα σύντομο σχόλιο και δύο ερωτήσεις για τον κύριο Πίτερ Ρέντινγκ. Πρώτον, Έχουμε μία αναφορά περίεργη ενό Γάλλου φαρμακοποιού που δεν μπορεί να λειτουργήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο φαρμακείο γιατί η Βρετανική νομοθεσία δεν το επιτρέπει. Το δικό σα το γραφείο μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την υπόθεση που είναι σαφής παραβίαση με το, προς τους, των κανόνων της Ένωσης. Δεύτερον, μπορεί να, προβλέψ, να προβλεφθεί ότι κάποια στιγμή θα υπογράψει και το Ηνωμένο Βασίλειο το χάρτη γιατί ε, ζήτησε εξαίρεση. Τέλος, πριν από λίγους μήνες άκουσα ότι ο Πρωθυπουργό Κάμερον εξετάζει τη δυνατότητα, το ενδεχόμενο, να μην εφαρμόσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασίλειο, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό σοκάρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι λέτε εσείς, πώς τα κρίνετε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν εδώ για να μας μιλήσουν. Και αυτό το οποίο μου φαίνεται ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως είπε στο τέλος ο Μπάτλερ, είναι το ότι δεν υπάρχει αυτή, υπάρχει αυτή η δυσκολία, δεν υπάρχει ενημέρωση πρώτα πρώτα επομένω. το ότι θα πρέπει να ξέρει ο Ευρωπαίος τα δικαιώματά του για μπορεί να το υπερασπιστεί. Επίσης, δεν υπάρχει κεντροκατευθυνόμενη ρύθμιση, όπως εξήγησε ο κύριος Μποντής. Γιατί στη Γαλλία, ας πούμε, υπάρχει μία και μόνο υπηρεσία και κατόπιν ε, υπάρχει ανακατεύθυνση του θέματος όπου πρέπει. Βεβαίως, ευτυχώς, που υπάρχει και αυτός ο χάρτης. γιατί ακριβώ τελικά προτεραιότητα έχει το θέμα της πράσπισης του Ευρωπαίου. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στο τι ισχύει για τον κάθε διαμεσολαβητή. Ο Πολωνός ας πούμε που ήρθε εδώ να μας μιλήσει έχει τρομερές αρμοδιότητες. Τρομερές εξουσίες. Και μπορεί επομένως να διορθώσει τα πράγματα όταν υπάρχει κάποια στρεβή ε, απόφαση. Θα πρέπει να διευκολυνθεί το έργο των διαμεσολαβητών και του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή επίση και να υπάρχει κάποιο είδου και το καθινόμενη ε, ρύθμιση, κάποια κεντρική υπηρεσία για τα δικαιώματα. Να, παράδειγμα, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. το πρόβλημα του Γιούγκεναμ στην ε, Γερμανία όσον αφορά το δίκαιο του διαζυγίου. Τι γίνεται λοιπόν όταν ο ένας από τους συζύγους είναι Γερμανός και ο άλλος δεν είναι. Συνέχεια προκύπτει αυτό το πρόβλημα. Μας έρχεται στην Επιτροπή. Εδώ και χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Και δεν επιλύεται το θέμα, γιατί δεν μπορεί η Επιτροπή των Αναφορών κάτι να κάνει. Μόνο κατευθύνσεις να δώσουμε, αντολισμό. Και πολλές φορές τους στέλνουμε κάπου που βρίσκουν βοήθεια. Τελικά όμως θα έπρεπε να γίνει ένας συντονισμός μεταξύ των διαμεσολαβητών. Και θα είχαμε πολύ καλύτερη κατάσταση. Επαναλαμβάνω επομένω. Γιατί υπάρχει τόση ποικιλία μεταξύ των αρμοδιοτήτων των διαμεσολαβητών. Υπάρχουν ούτε διαμεσολαβητές. Γίνεται όταν έχουμε κάποιο συντονισμό μεταξύ των μεσολαβητών. Και άλλη μια ερώτηση νομίζω υπήρχε από εδώ, από ένα άλλο μέρος. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που δεν παρακολούθησα όλη την ε, συνεδρίαση, αλλά θα ήθελα να προσθέσω στο σχόλιο σας. Έχουμε εδώ ε, ένα διμερές θέμα, ε, ε, ε, βάλατε θέμα διμερές μεταξύ ας πούμε Ισπανίας Ένωσης. Υπάρχουν κι άλλοι όμως και Γερμανοί και άλλοι πολίτες και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι ισπανικό μόνο το ζήτημα, αλλά πρόκειται για θέμα ευρωπαϊκό. Και θα ήθελα παρακαλώ αυτό να το σεβαστούμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και άλλη μια ερώτηση και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις. Μια τελευταία ερώτηση θα ακούσουμε τώρα. Ναι, ακόμα θα, θα μιλήσω γερμανικά, αφού έχουμε ακόμα τους διερμηνείς. Δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση προς τους διάφορους διαμεσολαβητές, οι συνηγόρους, οι εκπροσώπους εθνικών φορέων και ιδρυμάτων. Με ποιο τρόπο έχετε πρόσβαση στην κοινή γνώμη σε ποιο βαθμό την επιδιώκεται και σε ποιο βαθμό διαφοροποιείται μεταξύ επιμέρους περιπτώσεων καταγγελιών και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πληθώρα παρομοίων καταγγελιών. Πώς κοινοποιείται ας πούμε τα λάθη, τα κακό σκήμενα, ε, έχω υπόψη μου εδώ τον Αυστριακό διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει τακτική εκπομπή στην τηλεόραση και σε σταθμό παγκόσμιας εμβέλειας παρουσιάζει τα προβλήματα. Επίσης μια ερώτηση στον Πίτερ Ρέντινγκ. Για... Κύριε Ρέντινγκ, για εσάς. Σύντομη ερώτηση προς εσάς. Να τα πω στα αγγλικά. Ε, έχουμε το χαρτί θεμελιωδών δικαιωμάτων, έχουμε όμως την Ηνωμένο ε, Βασίλειο, την Πολωνία, ίσως και την Δημοκρατία της Τσεχίας, αν ε, δεχτούμε την τροποποίηση στη συνθήκη. Ε, αυτές οι τρεις χώρες έχουν ζητήσει εξαίρεση. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Ποια είναι η διαφορά που κάνει αυτή η εξαίρεση για τον κόσμο. Ωραία. Ο Ισπανός συνάδελφος τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την κυρία Άουκεν. Θέλω να πω ότι με ρώτησε μία σειρά πραγμάτων. Πρώτα-πρώτα ε, για το δικαϊκό σύστημα της χώρας, για το ότι είναι ε, ότι, ότι, ότι λειτουργεί με βραδίτητα και τι γίνεται με τους διαμεσολαβητές και για το... προσπαθούμε, κάτι να κάνουμε. Προσπαθεί, προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί. Ε, μιλάμε ο, για το ότι προσπαθούμε να, να παράσχουμε τις εγγύησεις που και έχουμε όλα, τα διάφορα επίπεδα δικαι, δικαιοσύνης και πρέπει να δούμε τα θέματα της ε, αρμοδιότητας του κάθε δικαστηρίου. Δεύτερον, ρωτήσατε εάν έχουμε αρκετή προστασία που παράσχουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους πολίτες. Γιατί από την Ισπανία λαμβάνεται πολλές καταγγελίες. Αυτό γίνεται. Ξέρετε και εγώ έχω συμμετάσχει στην Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου μας Τέσσερις θητείες έκανα στην, ε, στο, στη Βουλή αλλά και στη Γερουσία και όντως είχαμε πολλές αναφορές. Όμως υποθέτω ότι αυτές οι αναφορές στις οποίες αναφερθήκατε ε, έρχονται γιατί στην Ισπανία έχουμε πάρα πολλούς ξένους που έχουν αυτή τη δεύτερη κατοικία και διαμαρτύρονται για, το, για την κατάσταση που ισχύει αλλά έχουμε και τις άλλες περιπτώσεις καταχρήσεως δικαιωμάτων, υποθέτω ότι η νομοθεσία μας, οι φορείς που έχουμε, ποτέ δεν θα αρκούν. Όμως, είναι σημαντικές οι ρυθμίσεις που υπάρχουν. Και παραλαμβάνω, έρχονται εδώ τόσες without translation, without mic. Ah, and using the microphone. So please, Mr. Boudis, if you just want to, si vous voulez choisir. Non, no, it's working. Maintenant, ça marche. Et est-ce qu'il y a encore la traduction Si. Maintenant, ça fonctionne. Traduction. Oui. Muy brevemente, si me permite el presidente, yo creo que ya, ya funciona, ¿verdad? ¿No? A mí sí. ¿Me oyen? français.